Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την ακρόαση, την δημόσια ακρόαση για το θέμα άνθρακας και αέριο. Φίλοι ή εχθροί, θα ήθελα να ζητήσω από αυτούς οι οποίοι θα πάρουν μέρος να πάρουν τις θέσεις τους. Ίσως να δώσουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας για να Bene, Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω όλους όσους πάρουν το λόγο σε αυτήν την ακρόαση. Τους ευχαριστώ εξ ονόματος της Προεδρίας και της Επιτροπής μας που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας και θα πάρετε μέρος σε μια ακρόαση σημαντική λόγω του θέματός της σχετικά με την οργάνωση αυτής της ακρόασης. Έχετε το πρόγραμμα μπροστά σας. Δύο είναι τα τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά τους σπόρους και το δυναμικό άνθρακα και αερίου στην Ευρώπη. Το δεύτερο τμήμα αφορά τις λεγόμενες οικονομικές πλευρές και τις εκπομπές καυσαερίου ε, από το αέριο και τον άνθρακα και τις συνέπειες που θα έχουν στην μελλοντική ενεργειακή μας πολιτική. 12 και 30 κλείνει η γι' αυτό παρακαλώ να σεβαστείτε τον χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας ήδη καθορισμένο. Θα ήθελα λοιπόν για να ξεκινήσω να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος δεν θα ήθελα να ξεπεράσει παρακαλώ τα 10 λεπτά. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το φυσικό αέριο και το ο ή έχθρη. ή εχθροί. Η απάντησή μου σε αυτό θα ήταν ούτε ούτε μήτε μήτε ουδέ μηδέ. Τα ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο ή ο άνθρακας θα εξακολουθήσουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι τμήματα του ενεργειακού μείγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος αυτών των ορυκτών καυσίμων στο μέλλον και στην εσωτερική αγορά ενέργειας, όλα αυτά θα εξαρτηθούν πρώτα απ' όλα από τον τρόπο με τον οποίο τα ορυκτά αυτά καύσιμα θα αντιμετωπίσουν τις αντίστοιχες προκλήσεις και πώς επίσης αυτά τα ορυκτά καύσιμα θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις νέες ευκαιρίες οι οποίες έρχονται με την εσωτερική αγορά ενέργειας και τη συμπληρωσή της. Για να σας δώσω ένα πλαίσιο σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να ατενίσω την τωρινή κατάσταση στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συγγνώμη, άνθρακος και φυσικού αερίου. Τα τελευταία δύο χρόνια. Το μερίδιο του άνθρακα αντίθετα με αυτό του φυσικού αερίου, έχει αυξηθεί σε πολλούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο κύριος λόγος γι' αυτό είναι η τιμή του άνθρακα. Η τιμή του άνθρακα έχει μειωθεί σταθερά, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι χαμηλές τιμές άνθρακα οφείλονται κυρίως σε στον μεγάλο όγκο εισαγωγών και εδώ βλέπετε τι κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες επενδύουν ιδιαίτερα για την ε, εσωτερική αγορά στην εξόρυξη αερίου από σχιστόλιθους, σχιστολιθικούς ε, σχηματισμούς και εξάγουν ένα μεγάλο τμήμα του παραγωμένου από αυτούς άνθρακα στην, ε, στο διεθνή χώρο και στην ε, Ευρώπη. Έχουμε επίσης σημαντικές εισαγωγές από την Κολομβία και τη Ρωσία. Οι χαμηλές τιμές άνθρακα συμβάλλουν στο φαινόμενο αυτό μεγαλύτερης χρήσης του άνθρακα και μεγαλύτερου μεριδίου, μεριδίου στην παραγωγή του άνθρακα. Οι χαμηλές τιμές άνθρακα εξάλλου οφείλονται σε μεγάλο βαθμό και στην, και από την, και στην οικονομική κρίση. Αν ατενίσουμε από την άλλη μεριά το τομέα του φυσικού αερίου βλέπουμε ότι εκεί οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τον άνθρακα. Αυτό οφείλεται ιδιαίτερα στην ε, σύνδεση των μακροχρονίων συμβάσεων της τιμής του φυσικού αερίου με την τιμή του αργού πετρελαίου. Βλέπουμε μια τάση αναδιαπραγμάτευσης αυτών των συμβολέων και μιας αποσύνδεσης από αυτήν την μορφή Σύνδεση τιμή φυσικού αερίου και πετρελαίου, αλλά τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι παραπάνω από 50% αυτών των μακροχρονίων ε, συμβολέων έχουν αυτή τη σύνδεση. Επίσης, οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνονται. Τα φορτία φυσικού, υγροποιημένου φυσικού αερίου πηγαίνουν περισσότερο στην ασιατική αγορά, όπου οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες. Τέλος, οι χαμηλές τιμές άνθρακα στο σύστημα εμπορίας ETS έχουν υποσκάψει ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα των σταθμών παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο. Ω εκ τούτου, τουλάχιστον με την τωρινή συγκυρία, οι παραγωγοί ενέργειας προτιμούν τους ε, σταθμούς που λειτουργούν με καύση άνθρακα και που φαίνεται να είναι πιο κερδοφόροι από ό,τι αυτή του φυσικού αερίου. Αυτό είναι τωρινή βέβαια κατάσταση το κατά πόσο θα παραμείνουν αυτές οι συνθήκες και στο μέλλον, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Γιατί όπως είπα προηγουμένως όλα αυτά εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πώς το φυσικό αέριο και ο άνθρακας θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν ενώπιον τους και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν τις ανανεώσιμες ενέργειες να αναφέρω τώρα ορισμένε προκλήσεις και για το φυσικό αέριο και για τον άνθρακα, χωρίς να πω σε λεπτομέρειες, γιατί φαντάζομαι ότι οι λεπτομέρειες αυτές θα προκύψουν από τις παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων, των εκπροσώπων των διαφόρων τομέων και τη συζήτηση που θα επακολουθήσει. Για τον άνθρακα οι προκλήσεις είναι καταρχήν η συμμόρφωση με τους περιορισμούς για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Η μείωση εκπομπών επίση ορισμένων ρήπων που πρέπει να επιβληθεί για να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τις νέες αυτές προδιαγραφές θα χρειαστούν σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση πολλών από τους τωρινούς σταθμούς ενέργειας. Κάποιοι σταθμοί ενέργειας θα πρέπει επίσης να καταργηθούν για το, στο μέλλον. Θα δούμε λοιπόν στο μέλλον αν αυτή η τάση η οποία <clears throat> διαφαίνεται θα οδηγήσει σε τέτοιου είδους επενδύσεις για αναβάθμιση σταθμών παραγωγής ενέργειας με άνθρακα και ακόμα και κατασκευή νέων σταθμών που χρησιμοποιούν άνθρακα. Αν υπάρξει αυτή η τάση που θα οδηγήσει σε αναβάθμιση, ανακαίνιση και νέες κατασκευές, τότε ο τομέας αυτός του, της παραγωγής από άνθρακα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο συνολικός στόχος μείωσης της περιεκτικότητας σε άνθρακα. Και εδώ η Κομισιόν έχει προωθήσει την εξή λύση μέχρι τώρα, την ε, συγκράτηση και αποθήκευση του άνθρακα, του διοξίδιου του άνθρακος. Τα σχέδια λοιπόν CCS, συγκράτησης και αποθήκευσης, μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει ιδιαίτερα καρπούς, ήταν απογοητευτική η λειτουργία τους. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν θα μπορέσουν αυτά να ευδοκιμήσουμε. Θα είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε τεχνολογία αυτή, την τεχνολογία CCS, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ελκυστική σε εμπορικό και βιομηχανικό επίπεδο, ώστε και να υποστηρίξει την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα. Και η τελευταία πρόκληση που θέλω να αναφέρω για τον άνθρακα είναι το μέλλον του συστήματος ETS, εμπορίας εκπομπών, προς το παρόν. Υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές άνθρακα, <clears throat> όπως είπα και προηγουμένως. Και αυτό οδηγεί σε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της παραγωγής άνθρακα από φυσικό αέριο. Ποιο θα είναι το μέλλον όμως του συστήματος ETS. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε την προηγούμενη εβδομάδα την πρόταση της Κομισιόν για την οπισθοφόρτωση ε, στο σύστημα ETS με το να αλλάξουν οι ημερομηνίες δημοπρασίας πιστοποιητικών εκπομπών αριών του θερμοκηπίου, διοξιδίου του άνθρακος. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ETS δεν έχει μέλλον. Η συζήτηση αυτή πρέπει να ξαναξεκινήσει και ενδεχομένω η συζήτηση αυτή θα εστιάσει περισσότερο στη τομή ενός ανανεωμένου συστήματος ETS. Αν στραφώ τώρα στο φυσικό αέριο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η ανάγκη για μεγάλες επενδύσεις στην ε, παραγωγή και στην διασύνδεση έχουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο ισχύει ήδη για αυτές τις επενδύσεις. Και εδώ έχουμε κύριε, δύο κύριους μοχλούς πρόθεσης για τα θέματα αυτά. Καταρχήν ο κανονισμός για τις κατευθυντήριες γραμμές για διευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας και το δεύτερο στοιχείο, ο δεύτερος μοχλός ανάπτυξης είναι η διευκόλυνση Connecting Europe. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο αυτό το οποίο χρειαζόμαστε όμως τώρα είναι μια ταχεία εφαρμογή και του κανονισμού και τη, της διευκόνησης Connecting Europe. Η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί, ιδίω για το δεύτερο θέμα αυτό. Επεξεργαζόμαστε ένα κατάλογο πανευρωπαϊκό για σχέδια ευρωπαϊκού συμφέροντος Έχουμε πολλές, πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για προγράμματα υποδομών που αφορούν και την ε, παραγωγή ηλεκτρισμού και τη διανομή μάλλον ηλεκτρισμού και το τομέα φυσικού αερίου και όλα αυτά φαίνονται πάρα πολύ ελπιδοφόρα ότι μπορούμε με το Connecting Europe να προχωρήσουμε σε σημαντική πρόοδο για τα θέματα αυτά. Αλλά για το τομέα του φυσικού αερίου θα ήθελα εν κατακλείδη να αναφέρω και δύο περαιτέρω προκλήσεις. Η πρώτη από αυτές είναι το γεγονός ότι χρειάζονται νέοι πελάτες. Δεν μπορεί κανείς να ακολουθήσει τα τωρινά σενάρια. Πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη ενεργητικότητα στον τομέα αυτό. Το φυσικό αέριο πρέπει να εξεύρει νέους πελάτες είτε στον τομέα ε, της παραγωγής ηλεκτρισμού είτε σε άλλο τομέα είτε στις μεταφορές. Και χρειάζεται να ενισχυθεί ο σύνδεσμος παραγωγής ενέργειας και παραγωγής αερίου, μετατροπής ενέργειας σε φυσικό αέριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ανανεώσιμες ενέργειες που έχουν μια ακανόνιστη, ε, ένα ακανόνιστο προφίλ παραγωγής. Αν μπορούμε την ενέργεια που παράγεται λοιπόν να αποθηκεύσουμε υπό μορφή φυσικού αερίου, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τι ανανεώσιμε ενέργειε και να έχουμε μια καλύτερη προετοιμασία για το μέλλον. Να συνεχίσουμε όμω με τα τωρινά σενάρια, κατά τη δική μου άποψη, δεν θα ενισχύσει ιδιαίτερα τον τομέα του φυσικού αερίου. Εν κατακλείδη λοιπόν, για μένα δεν υπάρχει το θέμα αντιπαλότητος φιλίας ή νίκους μεταξύ φυσικού αερίου και άνθρακος και οι δύο πηγές αυτές είναι πολύ σημαντικές για το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, τουλάχιστον για το όρατο μέλλον. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες προκλήσεις που αν δεν αντιμετωπιστούν από τους αντίστοιχους τομείς, μπορεί αυτές οι προκλήσεις να τους αποσπάσουν την δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή την οποία κάνατε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και με σημεία για σκέψη. Θα δώσω το λόγο τώρα. Στη θέση της κυρίας Ολίβα θα μιλήσει ο Μάρτσιν Λέβενστάιν Θα ήθελα παρακαλώ να μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά. για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέγομαι Μάρτσιν Λεβενστάιν, εκπροσωπώ την πολωνική επιχείρηση Θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη από πλευρά της κυρίας Πετρόσκα Ολίβα, η οποία δεν είναι σε θέση να είναι μαζί μας σήμερα. Και θα συνεχίσω την ομιλία μου στα πολωνικά, έτσι ώστε να εκφραστώ καλύτερα και συντομότερα. Και ευχαριστώ για τις υπηρεσίες διευμηνίας που παρέχετε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, το φυσικό αέριο είναι ένα, μια, ένα υλικό το οποίο βρίσκεται σε όλο τον κόσμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα σπίτια, από τα νοικοκυριά και για θέρμανση αλλά και από τη βιομηχανία μεταφορών. Όταν τίθεται το θέμα λοιπόν πού συναντώνται ο άνθρακας με το αέριο, τότε η απάντηση είναι ο τομέας της ενέργειας. Στην αγορά ενέργειας και στα πλαίσια της αγοράς ενέργειας θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε αν είναι φίλοι ή εχθροί. Δεν είναι ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Είναι απλοί ανταγωνιστές. Από τη μία Υπάρχει μια κρίση. Από την άλλη θα πρέπει να αυξήσουμε την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τη ζήτηση και να εισάγουμε επίσης με αυξανόμενο συνεχώς τρόπο και τις ανανεώσιμες πηγές. Τώρα κάποιοι πρώτοι υπολογισμοί, τους οποίους έχουν κάνει εμπειρογνώμονες σχετικά με τον ανταγωνισμό το φυσικό αέριο φαίνεται να πηγαίνει καλύτερα από τον άνθρακα. Το ανταγωνιστικό φαίνεται ότι είναι πιο, το φυσικό αέριο είναι πιο ανταγωνιστικό από άλλες ύλε και πράγματι πολλαπλασιάζονται τα σημεία διασύνδεσης και τα σημεία αποθήκευσης σε διάφορα σημεία της Ευρώπης. Και στη Βόρεια Θάλασσα και στη Μαύρη Θάλασσα και στο ανατολικό τμήμα της Μεσογειακής Λεκάνης έχουν ανακαλυφθεί πρόσφατα νέες ποσότητες φυσικού αερίου. Η απελευθέρωση των αγορών επίσης ε, ε, βοηθάει όπως επίσης και οι κοινοτικές ρυθμίσεις για αυστηρές περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε αυτό το ευρύτερο λοιπόν περιβάλλον θα έλεγε κανείς ότι το φυσικό αέριο θα πήγαινε πάρα πολύ καλά τουλάχιστον σε σχέση με τα άλλα ορυκτά καύσιμα. Υπάρχουν βασικά τρεις κατηγορίες πλεονεκτημάτων του φυσικού αερίου σε σχέση με άλλα ορυκτά καύσιμα. Έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, έχει σχέση επίσης με την ευελιξία. Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιείται πιο εύκολα και τέλος να μιλήσουμε λίγο για τον οικονομικό τομέα, για τις επενδύσεις, για το περιβάλλον πρώτα. Οι εκπομπές του φυσικού διοξιδίου του άνθρακα είναι χαμηλότερες στην περίπτωση του άνθρακα από του φυσικού αερίου, συγγνώμη, από ότι άλλες πρώτες ύλες. Αλλά και στον τομέα των θιούχων έχουμε χαμηλότερες εκπομπές. Ταυτόχρονα ε, το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να υπάρξει συμπαραγωγή ενέργειας από διαφορετικές πηγές. Η ευελιξία λοιπόν είναι κάτι που χαρακτηρίζει το φυσικό αέριο. Η ευελιξία στο φυσικό αέριο είναι πάρα πολύ υψηλή. Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική πηγή για τις ανανεώσιμες πηγές ή καλύτερα για την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες. Το φυσικό αέριο μπορεί να αποθηκευθεί αρκετά εύκολα έτσι ώστε να καλύψουμε πιθανές διακυμάνσεις της ζήτησης. Η παραγωγή ενέργειας από το φυσικό αέριο είναι αντικείμενο ρύθμισης μέσα σε λίγα λεπτά και αν τυχόν αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και επειδή ακριβώς οι ανανεώσιμες πηγές εξαρτώνται από, το, από τις φυσικές συνθήκες, από τις κλιματικές συνθήκες και ποικίλουν σε σχέση με το μέγεθος της παραγωγής, μπορεί το φυσικό αέριο να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Και μπορεί επίσης το φυσικό αέριο να χρησιμοποιηθεί είτε σε ευρεία κλίμακα είτε σε περιορισμένη κλίμακα ανάλογα με τη διακύμανση των αναγκών. Ε, παρενθετικά να πω εδώ ότι το θέμα της αποθήκευσης της ε, ενέργειας είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την τεχνολογία. Ε, σας είπα τις δυνατότητες που παρουσιάζει σε σχέση με άλλες πρώτες ύλες το φυσικό αέριο. Και σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές θα υπάρξει η δυνατότητα αυτή στο μέλλον. Τώρα, ε, να μιλήσω για τον τομέα των επενδύσεων, τον οικονομικό τομέα και τα πλεονεκτήματα τις οποίες παρουσιάζει ε, τα οποία παρουσιάζει το φυσικό αέριο σε σχέση με άλλες πρώτες ύλες. Υπάρχει δυνατότητα σχετικά εύκολη και γρηγορότερη δημιουργία αγωγών φυσικού αερίου από ό,τι για άλλες πρώτες ύλες. Αυτά είναι λοιπόν τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου. Παρ' όλα αυτά δεν εκμεταλλευόμεθα πλήρως τις δυνατότητες που παρουσιάζει το φυσικό αέριο γιατί υπάρχει ένα βασικό θέμα. Ποιο είναι αυτό, η τιμή. Η τιμή είναι ένα εμπόδιο, είναι τροχοπέδι στην ανάπτυξη του τομέα του φυσικού αερίου. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται έντονα σήμερα. Έχει δύο βασικούς ανταγωνιστές στο φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές που προστατεύονται από επιδοτήσεις και από την άλλη τον άνθρακα. Ο άνθρακας θα έλεγα λειτουργεί πλεονεκτικά λόγω της χαμηλής του τιμής. Και έτσι λοιπόν πιέζεται το φυσικό αέριο. Η ζήτηση για τον άνθρακα αυξάνεται ενώ η ζήτηση για το αέριο μειώνεται. 8% αυξήθηκε πέρυσι η ζήτηση του ε, άνθρακα ενώ 17% μειώθηκε η ανάγκη για φυσικό αέριο. Σε άλλες ε, περιοχές που χρησιμοποιείται το αέριο από σχιστολιθικές πηγές, εκεί τα πράγματα διαφέρουν. Οι μη συμβατικές αυτές μορφές παραγωγής δηλαδή έχουν οδηγήσει στις Ηνωμένε Πολιτείες σαν παράδειγμα σε μια ισορροπία ανάμεσα στις διακυμάνσεις της συζήτηση του φυσικού αερίου και του άνθρακα. Βλέπουμε όμως ότι έχουμε στις Ηνωμένε Πολιτείες και με νέες βιομηχανίες οι οποίες είχαν φύγει τα τελευταία χρόνια και επανέρχονται λόγω της διαθεσιμότητας φυσικού αερίου από σχιστολιθικές ε, ε, πηγές. Αυτό είναι θα έλεγα ε, μια δυνατότητα που στην Ευρώπη ακόμα δεν έχουμε. Οι πολιτικές των κρατών μελών απέναντι στην παραγωγή ενέργειας από σχιστολίθους ε, είναι κάτι το οποίο ε, βρίσκεται σε ε, μια πρώτη φάση, πρώιμη φάση. Κάποιες χώρες έχουν εγκαταλείψει τις δυνατότητες αυτές και αυτό είναι κρίμα γιατί ακόμα και αν δεχθούμε κάποιες πολύ συντηρητικές προβλέψεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι το αέριο από σχιστολιθικές πηγές θα μας δώσει 30 χρόνια ενεργειακής ανεξαρτησίας στην Ευρώπη, αν πράγματι εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες. Εμείς στην Πολωνία θέλουμε να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες αυτές. Πιστεύουμε ότι έχουμε την δυνατότητα ε, για γρήγορη εκμετάλλευση και εξαγωγή αερίου ιδιαίτερα στην κεντρική και την βόρεια Πολωνία, στην περιοχή της Λεκάνης της Βαλτικής όπως την ονομάζουμε. Θέλουμε εμείς να προχωρήσουμε σε 13 με 15 ε, προοπτικές εξόριξης στην περιοχή. Αυτό θα αυξήσει την παροχή φυσικά του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά και αυτό θα μπορέσει να αντικαταστήσει και αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει σήμερα. E, e, e, το θέμα της σύνδεσης με την τιμή του πετρελαίου, της τιμής ε, του φυσικού αερίου. Κάτι το οποίο ορίζει πολλές τιμές όπως ε, και οι ε, τιμές του ηλεκτρισμού. Ξέρετε ότι βέβαια οι τιμές του πετρελαίου ορίζονται από γεωστρατηγικά κριτήρια και γι' αυτό ακριβώς είναι εντελώς ε, λάθος και αρνητική η διασύνδεση των τιμών των δύο πρώτων υλών. Πιστεύουμε ότι μέσω της εκμετάλλευσης των σχιστολιθικών πηγών θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε και να περάσουμε σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών. Αυτό βέβαια απαιτεί περαιτέρω μέτρα και σε επίπεδο διακανονιστικό και σε επίπεδο πληροφόρησης και ενημέρωσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το τι κάνουν φυσικά οι ανταγωνιστές μας. Όταν μάλιστα λαμβάνουμε υπόψη τα χρέη, τα δημόσια, τα υψηλότατα τα οποία χαρακτηρίζουν τις ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε τι γίνεται στην ΣΥΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στο Μεξικό και στην Νότια Αφρική αλλά και στην ίδια την Κίνα. Μου ζήτησαν να συντομεύσω οι οργανωτές γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Λοιπόν θα τελειώσουμε κάποιες γενικές σκέψεις. Παρακολουθώ προσεκτικά τις συναντήσεις που έχει ο τομέας, ε, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Συζητάμε λοιπόν για το μέλλον του φυσικού αερίου, το οποίο όμως βιώνουμε στην παρούσα φάση. Κοιτάξτε δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσουν και οι άλλοι να μιλήσουν. Καταφέρατε όμως να μας δώσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ο επόμενος ομιλητής Μάρακ Γέλινε και για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να σας δώσω μια πρακτική περισσότερο επισκόπηση κατευθείαν από την ε, βιομηχανία της, ε, του φυσικού αερίου. Εγώ προσωπώ τον μεγαλύτερο ε, παραγωγό ε, άνθρακα, επομένως ε, νομίζω ότι έχω μια καλή εικόνα της κατάστασης. Εμείς απασχολούμε περίπου 17.000 εργαζομένους σε τέσσερις χώρες και ε, παράγουμε 10 ε, δισεκατομμύρια τόνους ε, άνθρακα συνολικά. Επόμενη διαφάνεια. Ας εξετάσουμε τι σημαίνει το. Ο άνθρακας σε παγκόσμιο πλαίσιο είναι, βρίσκεται άφθονο στη φύση. Περίπου το 50% των παγκοσμίων αποθεμάτων ενέργειας βρίσκονται ε, σε άνθρακα και έχει καταναμηθεί μάλλον ε, ε, ισόποσα σε όλο τον κόσμο, σε χώρες που είναι ασφαλείς και με κράτος δικαίου, δηλαδή δεν βρίσκεται μόνο σε χώρες όπου υπάρχουν επικίνδυνες καταστάσεις όπως συμβαίνει με το πετρέλαιο. Είναι η μεγαλύτερη πηγή καυσίμου σήμερα. Επόμενη διαφάνεια. Να επικεντρωθούμε ε, στην κατάσταση στην Ευρώπη σε ό,τι τον άνθρακα. Περίπου ένα τέταρτο της ευρωπαϊκής ενέργειας ε, προέρχεται από τον άνθρακα. Είναι εξαιρετικά σημαντική πηγή λοιπόν και σίγουρα αυτό θα ε, εξελιχθεί στο μέλλον και θεωρώ ότι κάποια στιγμή η Ευρώπη και ο κόσμος θα περάσει σε μία, ε, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όμως θα μας πάρει αρκετά χρόνια. Και από τον τίτλο και όλες τη σημερινή ακροασίε, μπορώ να σα πω ότι ο άνθρακα δεν χρειάζεται να είναι εχθρό, μπορεί να είναι ένας σύμμαχο. Ένα στοιχείο που θα μας επιτρέψει ε, να κινηθούμε ε, προς έναν οικονομικά αποδοτικό και, και εταιρικά υπεύθυνο τρόπο μετάβασης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο άνθρακα αποτελεί μεγάλο τμήμα τη ευρωπαϊκή αγορά ενέργεια, 25%. Και αν δείτε τα αποθέματα ε, εκτό των ορυκτών καυσίμων, περίπου 80% των ε, αποθεμάτων ε, των ορυκτών αποθεμάτων ενέργειας βρίσκονται σε άνθρακα. Όμως εκπροσωπούμε, συγγνώμη, εισάγουμε τεράστιες ποσότητες άνθρακα και αυτό σίγουρα είναι παράγοντας και των παγκόσμιων τιμών άνθρακα, όμως είναι και ένα ερώτημα. Γιατί εισάγουμε όλων αυτών των άνθρακα, άλλες χώρες ε, δημιουργούν την απασχόληση και τον πλούτο. Η Ευρώπη, είμαι πεπισμένος ότι θα μεταβεί ε, σε μεγάλο βαθμό ή ακόμα και πλήρω ε, ε, στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ένα τέτοιο ενεργειακό μείγμα, αλλά αυτό θα μα πάρει δεκαετίε. Και για να σας τα πω και ξεκάθαρα, σίγουρα ο άνθρακας έχει και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εμείς και ως ε, βιομηχανία άνθρακα και ο κλάδος γενικότερα θα πρέπει να τα πάμε καλύτερα. Και θυμάμαι πώς ήταν και τα βορειοδυτικά ε, σημεία της ε, χώρας μου πριν από 20 χρόνια. Καμία σχέση ε, με τη σημερινή κατάσταση. Όμως και πάλι πρέπει να αλλάξουμε, να γίνει ο άνθρακας πιο καθαρός. Αλλά και πάλι υπάρχει σε αυθονία, είναι οικονομικά αποδοτικός πόρος και πολύ καλά θα κάνουμε να τον αξιοποιήσουμε. Και βεβαίω και οι ρυθμιστικέ αρχέ, οι κυβερνήσει πρέπει να ασκούν πιέσει στου κλάδου τη βιομηχανία, για να γίνουν πιο καθαροί, αλλά πάντα βάσει της λογικής. Προχωρούμε. Ο άνθρακας είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της μετάβασης αυτή τη στιγμή. Αν δείτε ε, το γερμανικό ενεργειακό μείγμα σήμερα πάνω από 5.000 ε, ε, ε ε, της ε, ικανότητας άνθρακα θα ξεκινήσει να αξιοποιείται ε, φέτος στη Γερμανία. Και υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες, μεγαλύτερη ικανότητα η οποία παραγγέλνεται αυτή τη στιγμή. Και η Γερμανία κάνει μια πολύ σημαντική μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρακας παραμένει ο πιο οικονομικά αποδοτικός ε, πόρος και δρόμος μετάβασης προς ε, τον ενεργειακό μείγμα. Επομένω, ο άνθρακας είναι εδώ και θα παραμείνει για αρκετά χρόνια. Επομένω, ε, θα πρέπει να δούμε αν θα αξιοποιήσουμε εμεί αυτή την ευκαιρία για να αυξήσουμε την απασχόληση ή αν θα δώσουμε σε άλλους φορείς τη δυνατότητα να το πράξουν. Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα είναι πολύ σημαντική ε, για μας ε, στη βαριά βιομηχανία Και το χαμηλό κόστος της ενέργειας, ή τουλάχιστον το διαχειρίσιμο κόστος της ενέργειας, είναι σημαντικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας. Ο συνάδελφος ε, προηγουμένως ανέφερε τις συνέπειες της λεγόμενης επανάστασης του σχιστολιθικού αερίου στις ΗΠΑ. Γιατί συνέβη αυτό, και στη Βόρεια Αμερική ε, εν γέννη. αυτό συμβαίνει γιατί παρέχει φθηνή ενέργεια. Και αυτό χρειαζόμαστε. Έχουμε, έχουμε φθηνή ενέργεια μέσα στα ευρωπαϊκά σύνορα. Γιατί δεν ε, βασιζόμαστε περισσότερο σε αυτήν λοιπόν. Είναι ένα καλό ερώτημα. Επίσης η μετάβαση προς ε, τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, ακόμα και στο σύνολο του ενεργειακού μείγματο, απαιτεί σημαντικέ επενδύσει. Ποιο θα τι αναλάβει. Πρέπει να δημιουργηθεί πλούτος που θα δημιουργηθεί από μια ανανεωμένη, νέα, καινούργια και αναζωογονημένη ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία, η οποία πρέπει να βασιστεί ε, σε αηφόρο ε, ενέργεια από με χαμηλό κόστος. Το σημείο του γονισμού ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδίω να εξετάσουμε και την κεντρική Ευρώπη, που προέρχομαι και εγώ ίδιο. Δύο στοιχεία έχω να αναφέρω εδώ. Πρώτον, ε, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, τη κεντρική Ευρώπη μάλλον, καθώ και η βιομηχανία τη κεντρική Ευρώπη ε, συγκριτικά πληρώνουν ε, μεγαλύτερο μερίδιο ε, του εισοδήματό του για την ενέργεια σε σχέση με τον μέσο όρο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η βιομηχανία εν γέννη και ο άνθρακας συγκεκριμένα απασχολούν ε, μεγάλο αριθμό εργαζομένων και στην Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη. Πολύ σημαντικές αυτές οι θέσεις απασχόλησης ε, στις οικονομίες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδίως ε, υπό το φως της σημερινής ύφεσης. Για παράδειγμα, το τμήμα της Ευρώπης που μας απασχολεί, το σύστημα, ε, η περιοχή της ε, Μοραβίας είναι η μεγαλύτερη περιοχή ε, στην Ευρώπη από πλευρά βιομηχανικής απασχόλησης. Περίπου 36% των ε, θέσεων απασχόλησης στον, στην περιοχή όπου δραστηριοποιούμεθα αφορούν τη βιομηχανία. Δύο φορές μεγαλύτερος αριθμός από το μέσο όρο της Ευρώπης. Επομένως, η ανταγωνιστικότητα είναι κρίσιμη σημασία για μα και θα δυσκολευτούμε να τη διατηρήσουμε αυτήν την ανταγωνιστικότητα αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να βασιστούμε μεταξύ άλλων ε, σε ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας ή ενεργειακών πόρων. Και παρεμπιπτόντω, γιατί υπάρχει αυτή η βιομηχανία σε αυτή την περιοχή, στη Μοραβία Σιλασία. Όχι επειδή είναι ε, φθηνέ θέσει απασχόληση. Υπάρχει εκεί εδώ και 200 χρόνια, επειδή υπάρχει άνθρακα στο υπέδαφο. Γι' αυτό και υπάρχει χαλιβουργία ε, στην Τσεχία και ε, στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό και η Τσεχία και η Σλοβακία είναι ε, ηγετικέ δυνάμει ε, στην ε, βιομηχανική παραγωγή ε, κατά κεφαλήν. Αν δείτε, τους, αν μιλήσετε στους πελάτες μας, οι χαλιβουργικές επιχειρήσεις, και εγώ συναντήθηκα προσφάτως μαζί τους, θα σας πούν όλοι ένα πράγμα, το εξής. Το μέλλον της, της κεντρικής Ευρώπης διασφαλίζεται επειδή υπάρχει άνθρακας. Αν δεν υπήρχε ο άνθρακα, όλε αυτέ οι βιομηχανίε δεν θα βρίσκονταν εκεί. Είναι λοιπόν κρίσιμη σημασία για την οικονομική μεγέθυνση τη Κεντρική Ευρώπη και για την απασχόληση στην περιοχή. Κλείνοντα λοιπόν. Να σας πω ότι θεωρώ ότι κάποια στιγμή η Ευρώπη θα ε, μεταβεί προς ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα είναι πιο εύκολο και οικονομικά αποδοτικό να το πράξει αν ε, βασιστεί σε οικονομικά αποδοτική πηγή ενέργειας, ε, που είναι ο άνθρακας, ε, που βρίσκεται σε αυθονία στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να παράσχει ε, απασχόληση στην Τσεχία, στην Πολωνία και άλλες χώρες και να δημιουργήσει πλούτο που θα χρηματοδοτήσει αυτή τη μετάβαση προς τις ανάσχομες πηγές ενέργειας, εν μέρη ή και στο σύνολο του ενεργειακού μείγματος. Και κλείνοντα μια προσωπική αναφορά, δεν μίλησα εδώ τόσο ε, για συγκεκριμένες, συγκεκριμένους όρους ε, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Βεβαίως και ο άνθρακας έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις και πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να γίνουμε πιο καθαροί, αν και υπάρχει πρόοδος. Ε, εμένα με εκπλήσει τόσο πολύ ε, το γεγονός ότι η ζωή στην γη ε, διατηρήθηκε για δισεκατομμύρια χρόνια μόνο με την ηλιακή ενέργεια και ε, μετά υπήρξε βέβαια βιομηχανική επανάσταση, αλλά θα φτάσουμε στον στόχο που θέλουμε αν βασιστούμε στους πόρους που βρίσκονται σε αυθονία γύρω μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους, τους οποίους να ζητήσω να μην μιλήσουν πάνω από δύο λεπτά, για να επιτραπεί στους ομιλητές μας να απαντήσουν. Ο κύριος Πρόντι έχει ζητήσει το λόγο. penso che non ci sia conflitto ε, ε, Νομίζω ότι το φυσικό αέριο είναι πραγματικά μια πολύ ευέλικτη ε, πηγή ενέργειας με προοπτικές υψηλότατης αποδοτικότητας ακόμα και σε επίπεδο χαμηλής χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλες μορφές σε επίπεδα πάντα χαμηλών ποσοτήτων παραγωγής να συνδυαστεί με άλλες ε, πρώτες ύλες, θα έλεγα, παραγωγής ενέργειας με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Ο άνθρακας φυσικά και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις προοπτικές που έχουμε. Νομίζω ότι θα ήταν λανθασμένο να βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τώρα το φυσικό αέριο, θα πρέπει, το, τον άνθρακα. Θα πρέπει να τον μετατρέπουμε σε φυσικό αέριο με αποδοτικό τρόπο και έτσι να έχουμε το φυσικό αέριο εύκολα χρησιμοποιήσιμο για την ταχύτατη παραγωγή υψηλών επιπέδων με αποδοτικότητα άνω του 50% και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και με παραγωγή σε υψηλή θερμοκρασία και για τη μέθοδο της παραγωγής αερίου. Certamente eh, il problema rimane della anidride carbonica, però eh, io credo che eh, eh, accanto al carbone bisogna considerare eh, la biomassa in particolare. Και με χαμηλές, εν πάση περιπτώσει, παραγωγές διοξιδίου του άνθρακα, σαν παράδειγμα η παραγωγή αυτή από πλευράς ε, των δασικών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων μπορεί να δώσει το 1 τρίτο των αναγκών σε φυσικό αέριο για μια χώρα σαν την Ιταλία. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να έχουμε λοιπόν από τη βιομάζα. Το θέμα είναι τον άνθρακα να μην τον κάψουμε αλλά να τον μετατρέψουμε σε φυσικό αέριο και να χρησιμοποιούμε τον ατμό που παράγεται σε υψηλή θερμοκρασία για να μην υπάρχει παραγωγή αζότου που θα δημιουργήσει άλλες δυσκολίες στα πλαίσια του καθαρισμού του διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει λοιπόν να διαμορφώσουμε εκ νέου την αρχιτεκτονική παραγωγής μας έτσι ώστε η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί να αντιμετωπιστεί σωστά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέλμερ έχει στήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για την ενεργειακή πολιτική μιλάμε για ένα τρίγωνο που περιέχει τρεις στόχους. Θέλουμε βιωσιμότητα, ασφάλεια εφοδιασμού και πρόσβαση προσιτή τιμή ενέργειας για να υποστηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα. Αλλά συμπεριφερόμαστε σαν το μόνο πράγμα που να μετράει είναι η βιωσιμότητα μέσα σε εισαγωγικά και δεν δίνουμε έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την προσιτή τιμή ενέργειας. Δεν μας νοιάζει η ασφάλεια εφοδιασμού. Δίνουμε πολλά λεφτά στι ανανεώσιμε ενέργειε, αλλά δεν δίνουν αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τη Γερμανία, όπου ήταν τεράστιε οι δαπάνε και οι επενδύσει στην ανανεώσιμη ενέργεια και παρόλα αυτά φτιάχνουν 25 νέου σταθμού <clears throat> παραγωγή από άνθρακα ενέργεια και αυξάνουν οι εκπομπέ του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταγωνιστεί με άλλε περιοχέ του κόσμου. Η Αμερική έχει το συστολιστικό αέριο από μεγάλο βάθο και περνάει μια αναγέννηση στο βιομηχανικό τομέα η Νέα Κορέα και η, Ιαπωνία χρησιμοποιούν ε, επίσης ορυκτές πηγές και πηγαίνουν πολύ καλά. Εμεί χρησιμοποιούμε τις πιο ακριβές πηγές ενέργεια και αναρωτιόμαστε γιατί δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις μας να πάνε αλλού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είναι πιο χαμηλά και τα πρότυπα του περιβάλλοντος. Εμεί εξάγουμε τις βιομηχανίες μας, εξάγουμε τις επενδύσει μας, τις θέσεις απασχόλησης αλλά και τις εκπομπές μας. Γιατί ενώ εμείς στην Ευρώπη συγχαίρουμε τους εαυτούς μας γιατί οι δικές μας εκπομπές οξυδίου του άνθρακος μειώνονται ή συγκρατούνται, αυτές οι εκπομπές για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δείτε και τις εκπομπές που προέρχονται από τα εισαγόμενα καταναλωτικά αγαθά, τελικά αυξάνονται σημαντικά. Η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για περίπου 12% των συνολικών εκπομπών αερίου θερμοκηπίου από την Ευρώπη, αλλά 25% από τις συνολικές παγκόσμιες εκπομπές λόγω της κατανάλωσής μας. Όλο και περισσότερο είναι σαφές ότι οι μεγάλες μας επιδοτήσεις και δαπάνες για την ανανεώσιμη τεχνολογία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν σε οικονομικό επίπεδο. Η ανανεώσιμη ενέργεια δεν είναι οικονομικά βιώσιμη. Και θα πρότεινα στους συναδέλφους να κατανοήσουν ότι η ιδέα της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής είναι μια ιδέα η οποία και αυτή δεν ευσταθεί. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, ομιλητές. Πολυλογικά και πρακτικά τα όσα μας είπαν. Ο τίτλος ε, είναι ενδιαφέρον. Όμως Όλα αυτά συνδέονται με μια εντύπωση που υπάρχει στην κοινωνία ότι εξαιτία των περιβαλλοντικών ε, ε, ζητημάτων ε, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας είναι εχθροί και πρέπει να καταργηθούν. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα γιατί τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε χάρη στο αέριο και στον άνθρακα δεν είναι εχθροί. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι εχθρός ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει ε, να εξετάσουμε εδώ και ίσως να αλλάξουμε και τον τρόπο σκέψης μας. Για μένα είναι μάλλον αντιφατικό να μιλάμε για τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση ε, που έχουμε αντιμετωπίσει και πώς θα ξεφύγουμε από αυτή, πώς θα αυξήσουμε την απασχόληση, πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί και ταυτόχρονα να μην χρησιμοποιούμε πρώτα απ' όλα τους ε, πόρους που έχουμε στην Ευρώπη και αντί να χρησιμοποιούμε αυτούς τους πόρους, να ε, δαπανούμε τεράστια ποσά σε εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Το 2011 η Ευρώπη δαπάνησε 388 δις ε, ευρώ για την εισαγωγή ε, πετρελαίου και άλλων καυσίμων. 53% της μικτής κατανάλωσης ήταν προϊόν εισαγωγής. Και όπως αναφέρεται, έχουμε και φυσικό αέριο και άνθρακα σε αυθονία και δυσκολεύουμε ακόμα και τη δική μας βιομηχανία να αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους. Ε, επίσης, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την αδειοδότηση και πάλι υπάρχουν εμπόδια. Χρειαζόμαστε μια διαφορετική συμπεριφορά προς ε, την βαριά βιομηχανία ε, την οποία αντιμετωπίζουμε διαφορετικά από ε, τις ε, τεχνολογίες και τις βιομηχανίες της πληροφορικής. Εκεί είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί και, και είναι ευπρόσδεκτοι. Όμως όταν μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία πάντα είμαστε πολύ πιο καχύποπτοι και θεωρούμε ότι αν μπορούμε να τα εισάγουμε, εισάγουμε αυτούς τους σπόρους από αλλού, τότε εντάξει δεν θα επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Αν όμως το παράξουμε εμείς στην Ευρώπη, τότε πλήττουμε το περιβάλλον. Είναι ένα σφαιρικό, παγκόσμιο πρόβλημα και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί πρέπει να ακολουθήσουμε ε, και να αξιοποιήσουμε τους πόρους μας. Τουλάχιστον να βοηθήσουμε την βαριά βιομηχανία να δραστηριοποιηθεί όπως συμβαίνει αλλού. Η κυρία Εύτσογκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα σχόλιο για τη σύνθεσή μας. Λυπάμαι που βλέπω συνάδελφοι ότι οι συνάδελφοι που είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών δεν είναι παρόντες. Και πάρα πολλοί από τους συναδέλφους που είναι παρόντες δεν συμμετέχουν στις συζητήσεις που γίνονται για τις ανανεώσιμες πηγές και αυτό είναι πάρα πολύ λάθος. Όσο είμαστε μαζί, τα θέματα των ανανεώσιμων θα είναι μπροστά μας, τα θέματα του φυσικού αερίου και του άνθρακα θα είναι μπροστά μας, η πυρηνική ενέργεια θα είναι μπροστά μας. Καιρός ήταν νομίζω να γίνει ένα τέτοιο σχόλιο, αν και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Μία ερώτηση. Μπορείτε να μου πείτε τρία πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ένωση για τη βιομηχανία σας. Λεσέφε να σας αφήσει να κάνετε ό,τι θέλετε. Θέλετε να προχωρήσουμε σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Τι ακριβώς θέλετε. Αν έχετε τρεις ευχές και εμείς ήμασταν οι νεράιδες σας. Τι θα θέλατε να κάνουμε για σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Χίμπνερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Εγώ παρακολουθώ τις εκθέσεις μας για τα θέματα αυτά που, συμπερι... που περιστρέφονται γύρω από τα θέματα ε, ε, ενέργειας και έχω ερευνήσει και εγώ μέσω των συνεργατών μου σε διάφορες πηγές το φυσικό αέριο θα κρατήσει 30 με 50 χρόνια, το αέριο που σχιστολήθος 20 χρόνια και το, ο άνθρακας καμιά εκατοστή χρόνια. Χρειαζόμαστε τεχνολογίες εχμής αυτή τη στιγμή για να καλύψουμε την ενέργεια για περίοδους εχμής. Για τις ανανεώσιμες ενέργειες δεν έχουν εξευρεθεί οι λύσεις για αυτό το θέμα. Χρειαζόμαστε όμως και κρυανοτόμες λύσεις για, τον άνθρακα και το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να παρουσιάζονται ως ανταγωνιστικές αυτές τις πηγές Ορισμένοι από εμά υποστηρίζουμε τα ανανεώσιμε ενέργειε, άλλοι του, τον άνθρακα και άλλοι το φυσικό αέριο. Όλα αυτά είναι στοιχεία του ενεργειακού μείγματο τη Ευρώπη και πρέπει σε όλα αυτά τα συστατικά να υποστηρίξουμε την καινοτομία. Είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή μονάχα να επιδοτούμε την ηλιακή ή την αιωλική ενέργεια, τις ενεώσιμες ενέργειες. Αυτό είναι δια είναι στρέβλωση της ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ισότητα ανταγωνισμού. Θέλω να αναφερθώ στον ομιλητή που μίλησε για τον άνθρακα. Ποια είναι η κατάσταση της έρευνας για καινοτόμες τεχνολογίες που βασίζονται στον άνθρακα πέρα από τη συγκράτηση και από την Έχουμε κάποιες ε, νέες τεχνολογίες, ε, νανοτεχνολογίες κτλ. Κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τον άνθρακα στο ενεργειακό μας μείγμα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ λοιπόν για όλα τα στοιχεία τα οποία μας έδωσαν οι ομιλητές μας να αναφερθώ σε αυτό το οποίο τώρα μόλις είπε η κυρία Χέρτσοκ. Πράγματι πολλές φορές είμαστε ιδιαίτερα περιοριστικοί και ξεχωρίζουμε τις διαφορετικές πηγές ενέργειας τη μία από την άλλη, ενώ θα έπρεπε να έχουμε μια συνολική αντίληψη και να ασχοληθούμε από κοινού με όλες τις πηγές. Αν τις συνδυάσουμε με σωστό τρόπο θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την παραγωγή ενέργειας. Δεν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στο φυσικό αέριο, τον άνθρακα κτλ. Σχετικά με το φυσικό αέριο, γνωρίζουμε ότι ορισμένες ομάδες και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν σαν στόχο να μποϊκοτάρουν τις λεγόμενες μη παραδοσιακές ή μη συμβατικές εν πάση περιπτώσει πηγές φυσικού αερίου. Αν και το αέριο το οποίο παράγεται από σχιστολιθικές πηγές έχει διαφορετική σύνθεση από ότι άλλες παραδοσιακότερες μορφές ε, παραγωγής. Υπάρχουν ορισμένα πιλωτικά προγράμματα που έχουν ξεκινήσει στην Πολωνία, ιδιαίτερα στην Άνω Σιλεσία. Και αυτές οι πηγές που προέρχονται από αεριούχους ορίζοντες ε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Χρειάζεται λοιπόν μια συνολική αντιμετώπιση και όχι μια ανταγωνιστική αντιμετώπιση. Έχετε δίκιο γιατί μέσα σε μια πάρα πολύ μικρή χρονική περίοδο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν οι παραδόσεις μιας βιομηχανικής υπήρου. Μιλάμε για συνήθειες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 200 χρόνια. Η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη είναι διαφορετική από ότι η κατάσταση στην Πολωνία. Παρ' όλα αυτά έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε με τις απαιτήσει του Κιώτο για τη μείωση των εκπομπών. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια των συζητήσεων για την αλλαγή του ενεργειακού μίξ που χρησιμοποιούμε. Αυτή λοιπόν η αντιπαράθεση, αυτή η, η θέση εν αντιθέτω διαφορετικών πηγών ενέργειας δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα είναι χρήσιμο. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και πρέπει να μπορούμε να αλλάξουμε τις αποφάσεις μας ε, γρήγορα. Μια συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στα βιοκαύσιμα, μια συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στις εναλλακτικές πηγές, ε, μία στον άνθρακα κτλ. Ξαφνικά ε, κολλάμε σε ένα θέμα, επιδιώκουμε μόνο την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα και όλα αυτά γίνονται πλήρη έλλειψη ισορροπίας εις βάρος των επιχειρήσεων και τα θέματα των κινήτρων ανάλογα με το η μορφή της παραγωγής ενέργειας και αυτό είναι κάτι το οποίο αλλάζει συνέχεια. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λοιπόν τις δυνατότητες για γρήγορη απόκριση στις αλλαγές. Ένα επιπλέον σχόλιο. Η αιωλική, παραγωγή αιωλική ενέργειας δημιουργεί προβλήματα μεταφοράς Ξέρετε ότι ο άνεμος δεν είναι συνεχής, έτσι η παραγωγή από αιωλική ενέργεια, αιωλικής μάλλον ενέργειας είναι ασυνεχής, μία είναι ιδιαίτερα ισχυρή, μία στιγμή είναι ιδιαίτερα χαμηλή και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στα δίκτυα μεταφοράς. Τώρα, η οικονομική βιωσιμότητα... Ceny węgla, ceny Σχετικά με την αποθήκευση του άνθρακα, τα οικονομικά μοντέλα τα οποία υπάρχουν, ε, ποια είναι και τι θα πρέπει να κάνουμε στα πλαίσια και της κρίσης την οποία βιώνουμε. Κοιτάξτε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Μπορείτε παρακαλώ 4 με 5 λεπτά το πολύ. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσετε εσείς. Δεν μπορώ να εκπροσωπήσω βέβαια το βιομηχανικό το, τομέα, ε, εκπροσωπώ την Κομισιόν, αλλά ε, θα προτιμούσα ίσως, ίσως θα ήταν πιο καλό να ξεκινήσω για να επαναλάβω αυτά που είπανε πολλοί από τους ομιλητές. Κατανοώ αυτό που λέτε ότι δεν χρειαζόμαστε ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορετικών πηγών ενεργειών, χρειαζόμαστε μια συνολική προσέγγιση για να μπορέσουμε να φέρουμε από κοινού σε ένα κοινό μείγμα όλες τις πηγές ενέργειας που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει όμως να είμαστε ισοδίκαιοι και σε σχέση με τις πηγές αυτέ της ενέργειας. Όταν ακούω τον κύριο Χίπνο και τον κύριο Χέλμερ ότι οι ανανεώσιμες ενέργειες έχουν πολύ ψηλή επιδότηση. Μα για πόσο καιρό εμείς επιδοτούμε τον άνθρακα. Μόνο το 2018 σταματούν οι επενδύσεις για τον ανθρακικό τομέα ξεχνάμε τι θα κοστίσει στους Ευρωπαίους καταναλωτές αν αρχίσουμε να καταργούμε και να θέτουμε σε αχρηστία τους πυρηνικούς σταθμούς. Τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτά είναι ισοδίκια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις μορφές ενέργειας με τον ίδιο τρόπο και όχι να επιλέγουμε μονάχα αυτές που μας βολεύουν ως στόχους. Αν θέλουμε να έχουμε μια συνολική προσέγγιση και μια σωστή προσέγγιση στο ενεργειακό μείγμα στην Ευρώπη, που να βασίστε στις περιφερειακές δυνατότητες και ευκαιρίες. Θα πρέπει να συνδυάσουμε όλες αυτές τις πηγές σε μια εσωτερική αγορά με ιδιαίτερα διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα για κάθε χώρα. Αυτό πρέπει να προχωρήσουμε. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουμε. Το θέμα των επιδοτήσεων είναι ένα ζήτημα. Ένα άλλο ζήτημα βέβαια είναι το θέμα των προτύπων δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι υπάρχει το θέμα της βιωσιμότητας. Ναι, τα, οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας μπορεί να έχουν ένα πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά το θέμα της βιωσιμότητας <clears throat> και της αηφορίας. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή σχεδόν αυτόματα είναι ανανεώσιμες και αηφόρες, θα πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το φυσικό αέριο και τον άνθρακα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και αυτές οι μορφές ενέργειας ανταποκρίνονται στα περιβαλλοντικά μας πρότυπα και τα οποία έχουν θεσπιστεί για αποχρόντες λόγου. Και κύριε Χέλμερ, δεν μπορώ να καταλάβω πως λέτε ότι δεν είναι οικονομικά βιώσιμες οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Έχουν περάσει μια μακρά περίοδο βελτίωσης ήδη και υπάρχει ένα μέλλον για την οικονομικά βιώσιμη χρήση αυτών των μορφών ενέργειας. Αυτό που κάνουμε σε επίπεδο επιδοτήσεως ως Κομισιόν είναι θα εκδώσουμε μια ανακοίνωση όπου θα αναλύουμε όλα τα τωρινά συστήματα υποστήριξης και επιδοτήσεως για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Θα αναλύσουμε τον αντίκτυπο που έχουν αυτά τα συστήματα υποστήριξη για τις ανανεώσιμες ενέργειες στην εσωτερική αγορά ενέργειας και να κάνουμε και προτάσεις. Όλα αυτά όμως μέσα στο γενικό πλαίσιο ότι η Κομισιόν πιστεύει ότι υπάρχει ένα οικονομικά βιώσιμο μέλλον για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Τελευταία παρατήρηση για τον κύριο Πρόντι. Ναι, είναι εύστοχο αυτό που είπατε. Είπατε και αυτό είναι σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι καινοτόμε τεχνολογίε σε όλου του τομεί. Εσεί αναφερθήκατε ιδιαίτερα στον άνθρακα. Ίσως μπορεί να προκύψει περαιτέρω με μεγαλύτερε δυνατότητε σύζευξη των ε, ενεργειακών φορέων. Εγώ μίλησα για τι ανανεώσιμε και το φυσικό αέριο, εσεί μίλησατε για τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Θα πρέπει να υπάρχει η περιθώριο για έρευνα σε νέες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ, λέει πρώτος. Ο κύριος ε, Λεβενστάιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα απαντήσω στα πιο φιλικά εντός οικών ερωτήματα, που είναι και τα πιο εύκολα. Για την επιχείρησή μας θα ήταν σημαντικό να υπάρξει στήριξη. για να μπορέσουμε να διαρευνήσουμε και το μη συμβατικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Αυτό είναι σημαντικό. Και μετά αυτό το σύστημα στήριξη θα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Όπως και το σύστημα εμπορίας εκπομπών θα πρέπει να είναι προβλέψιμο, πρέπει να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Να είναι ένα επαρκέ σύστημα ε, με σκοπό την κάλυψη των ε, αναγκών ε, των φορέων, των εμπορευμένων. Γιατί αυτοί οι φορεί πρέπει να λάβουν αποφάσεις μακροπρόθεσμα με πολύ υψηλά ποσά. Και είναι δύσκολο να ε, πάρουμε αυτέ τι αποφάσει αν δεν γνωρίζουμε ακριβώ την κατάσταση. Μετά ε, δράτω με τι ευκαιρίε ε, για να σα πω το εξή. Ε, δεν... Ε, μιλώ για διασυνδέσεις, λέω ότι πρέπει να διερευνήσουμε περισσότερο για τη δέσμευση της ενέργειας, την αποθήκευση της ενέργειας. Αυτό είναι το σημείο κλειδί για το μέλλον και μπορεί να μας οδηγήσει ε, στην επιτυχία στην Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Θα ήταν ε, θετικό και για τις ε, για την οικονομία χαμηλής, χαμηλών εκπομπών άνθρακα Βεβαίω, ε, για το σχεστελιστικό ε, αέριο είναι μια πολλά υποσχόμενη ε, οικονομία, όμως υπάρχουν και προβλήματα γιατί με αυτούς τους λίθους που εξορίζονται είναι δύσκολη η παραγωγή ε, του φυσικού αερίου, γιατί υπάρχει το λεγόμενο gas reaction, αυτή η αντίδραση ε, κατά την οποία εκλείεται και το εξιδίο το άνθρακα. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο τόσο καλή ιδέα η παραγωγή αερίου με αυτόν τον τρόπο, γιατί το αέριο αυτό προκύπτει από χημική αντίδραση, που ούτε και αυτό είναι τόσο θετικό. Κάτι άλλο, σε ό,τι αφορά την παραγωγή αερίου, ε, θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το χρησιμοποιηθεί από τη χημική βιομηχανία. Ευχαριστούμε κύριο Τζελίνεκ. Thank you. I'll, just, I'll just quickly... Ο εγώ θα σταθώ τα ερωτήματα για τις νέες τεχνολογίες, το πώς μπορεί να μετατραπεί ο άνθρακας σε ενέργεια με νέες ε, τεχνολογίες. Υπάρχουν διάφορες ε, κατευθύνσεις ανάπτυξης στον τομέα αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι πολλά χρόνια από την ε, βιομηχανική ή εμπορική εκμετάλλευση. Εγώ δεν είμαι τεχνικός, είμαι οικονομικός εμπειρογνώμων και νομίζω ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι ακόμα ανταγωνιστικές, ως εκ τούτου, εμείς ως εταιρεία που χρησιμοποιεί τον άνθρακα μπορεί να αναπτύξει αυτές, μπορούμε να αναπτύξουμε αυτές τις τεχνολογίες σαν ε, χόμπι ουσιαστικά και όχι επειδή θεωρούμε ότι μπορούν να αποδώσουν καρπούς σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Και για τις τρεις ευχές, τις τρεις επιθυμίες που αναφέρατε προηγουμένως. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεστε δεν είναι να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών πηγών ενέργειας, απλώς χρειάζεται να υπάρξει μια αναλογική και λογική ε, αντιμετώπιση για να μπορέσουμε να περάσουμε το χάσμα το οποίο μας χωρίζει από ένα μέλλον ανανεώσιμης ενέργειας. Και επαναλαμβάνω και μερικά πράγματα που είπαν οι αδελφή μου. <clears throat> Χρειαζόμαστε σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Χρειαζόμαστε μια μακρο, μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση, μια μακρόπνο αντιμετώπιση. Αυτό το οποίο σίγουρα δεν χρειαζόμαστε είναι να μας βαραίνει το τεράστιο κόστος της ενέργειας, όπως είπα προηγουμένως και στην παρουσίασή μου. Ξέρω ότι δεν είναι μια συζήτηση για την ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά η Ευρώπη έχει να περάσει χαλεπούς καιρούς στο μέλλον. Και αν δεν, <clears throat> δεν καταλαβαίνετε ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εξωτερική βιομηχανία <clears throat> άνθρακα και η χαλιβουργία στην Ευρώπη, δεν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Η μόνη λύση για όλα αυτά είναι το να έχουμε ενέργεια σε προσιτή τιμή το μοναδίο κόστος του λεκτισμού θα αυξηθεί κατά 11% στο μέλλον, ενώ μειώνεται το κόστος του άνθρακα που πουλάμε κατά 10%. Όλα αυτά λοιπόν δεν βγάζουν νόημα. Έχουμε ένα σημαντικό λοιπόν πρόβλημα και εσείς έχετε τη δυνατότητα να βοηθήσετε την ευρωπαϊκή βιομηχανία να αντιμετωπίσει ένα αναπόφευκτο, μια αναπόφευκτη σειρά από δυσκολίες. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, ε, έπρεπε να γίνει αυτή η αναλλαγή στην Προεδρία. Σας ευχαριστώ για τις ομιλίες σας και ξεκινάμε τώρα την αλλαγή ανάμεσα στα δύο πάνελ. Θα πάρει το λόγο ο Μάρκους Τρίλινγκ και μετά ο τη.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 Δίνουμε λοιπόν το λόγο για 10 λεπτά στον, στον Μάρκου Τρίλινγκ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω και επίσης και του προηγούμενους ομιλητές γιατί κατέδειξαν το ρόλο του άνθρακα και του φυσικού αερίου για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακος και ανανεωσίμων ενεργειών. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι σε μακροπρόθεσμο επίπεδο οι επενδύσεις και η ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα θα πρέπει να φύγουν από τα ορυκτά καύσιμα και θα ήθελα για 10 λεπτά να αντιμετωπίσω λιγάκι τις οικονομικές συνέπειες της <clears throat> απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και να δούμε και ποιος είναι και ο ρόλος της δημόσιας χρηματοδότησης των δημοσίων τραπεζών για τα θέματα αυτά και θα εξετάσω επίσης το συνολικό πλαίσιο ενέργειας στον ορίζοντα του 2050 και την ανάγκη για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά θα καταλήξω στο συμπέρασμα ότι τολικές πολιτικές ε, χρηματοδότησης είναι μια στρέβλωση και πρέπει να σταματήσουν οι τράπεζες να υποστηρίζουν τα ε, ορυκτά καύσιμα. Εργαζόμαστε και σε συνεργασία με διεθνή χρηματοδοτικά ιδρύματα. Είμαστε λοιπόν ένα δίκτυο από μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται τα θέματα αυτά. Ο κύριος Κέλλη είπε σωστά ότι η Ευρώπη πουλάει τον πλούτο της στην ε, βιομηχανία ορυκτών καυσίμων. 53,8% της συνολικής ε, κατανάλωσης ενέργειας, 355 δισεκατομμύρια και οδηγεί αυτό σε ένα εμπορικό έλλειμμα 185 δισεκατομμύριων ευρώ. Αν δούμε τώρα την ανάγκη μετάβασης η οποία πρέπει να γίνει προς τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τη στρατηγική χαμηλής χρήσης άνθρακος. Και ένα slide πίσω παρακαλώ. και η λογική αυτή τη στατική χαμηλή χρήση άνθρακο είναι ότι πρέπει να μειώσουμε την επίπτωση στην κλιματική αλλαγή σε ένα λογικό επίπεδο. ένα πυλώνα αυτή τη στρατηγικής χαμηλή χρήση άνθρακο είναι ο ενεργειακό τομέα, ο οποίο θα πρέπει να απεξαρτηθεί τελείω από τη χρήση άνθρακα μέχρι το 2050. Ακούσαμε πόσο μεγάλη πρόκληση είναι αυτό από τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά αυτή είναι η χρονική στιγμή πού θα πρέπει να δημιουργηθεί η ενεργειακή υποδομή για το μέλλον. Μιλάμε για μια ενεργειακή υποδομή η οποία θα λειτουργήσει για, τα επόμενα, για τις επόμενες δεκαετίες. Οι επενδυτικές αποφάσεις λοιπόν του σήμερων θα διαμορφώσουν το ενεργειακό μείγμα του επόμενου μισού της, του αιώνα μας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, πρέπει να λάβουμε υπόψη για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. 80% όλων των εκπομπών που επιτρέπονται μέχρι το 2035 θα είναι δεδομένες λόγω των τωρινών σταθμών ενέργειας ε, των ε, εργοστασίων, κτηρίων κτλ. Αν συνεχίσουμε λοιπόν να αναπτύσσουμε την παραγωγή άνθρακα και τη χρήση άνθρακα, ε, δεν θα μπορούμε να έχουμε άλλες δημιουργίες υποδομών που παράγουν αέρια του θερμοκηπίου. Και πού βρισκόμαστε με τη διαδικασία αυτή μείωσης της ε, χρήσης άνθρακα από τις οικονομίες μας. Η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα είπε και ήταν κάπω απεσιόδοξη δεν υπάρχει πρόοδο, είπε, για την καθαρή ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο είναι βρώμικη ενέργεια τώρα, τόσο βρώμικη όσο πριν από 30 χρόνια. Ζητεί να υπάρξει μια επιτάχυνση της μετάβασης από τις ακάθαρτες πηγές, δηλαδή τα ορυκτά καύσιμα και επίσης να καταργηθούν σταδιακά οι επιδοτήσει στα ορυκτά καύσιμα. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Μιλάμε για την σχέση κόστους και ωφέλους, πόσο φτηνά είναι ορισμένα ορυκτά καύσιμα Προχωρούμε. Η τιμή του άνθρακα τώρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί υπάρχει τεράστιο κόστος υγείας το οποίο συνδέεται με την καύση ολικτών καυσίμων. Υπάρχει μια έρευνα που λέει 40 δισεκατομμύρια το χρόνο, 8 δισεκατομμύρια σε επίπεδο υγειονομικού κόστους στην Πολωνία το χρόνο, όλα αυτά μπορεί να τα διαμφισβητήσει κανείς, αλλά η καύση ορυκτών καυσίμων έχει πολλές πτυχές κόστους που δεν τιμολογούνται στο τωρινό σύστημα. Και επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα που αναφέρθηκε προηγουμένως, οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα. Και εδώ και παγκοσμία υπάρχει μια σαφής αντιμετώπιση που λέει ότι πρέπει να υπάρξει για τις επόμενες δεκαετίες κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα. Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν το οικονομικό όφελος το οποίο μπορεί να προκύψει σε ό,τι αφορά τις εκπομπές, σε ό,τι αφορά την ζήτηση για ενέργεια. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να σταματήσουν να σταματήσει η χρήση των ορικτών καυσίμων και το 2007 ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταματήσουν οι δημόσιες τράπεζες επενδύσεων και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα να σταματήσουν να υποστηρίζουν σχέδια που εμπλέκουν ορυκτά καύσιμα. Και μια πρόσφατη μελέτη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που δεν φαίνεται πάντα να είναι ο καλύτερος συνεργάτης των ΜΚΟ, μιλάει για, δι... για στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας και ότι οι τιμές ενέργειας να ανταραπλούν το πραγματικό κόστος. Είναι πολύ σαφές. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αυτή τη μελέτη του Απριλίου 2013 λέει ότι έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε οικονομικό επίπεδο οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα οδηγούν σε ανισομέρειες στον δημοσιονομικό τομέα, εμποδίζουν σημαντικές επενδύσεις στο δημόσιο τομέα, μειώνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και οδηγούν σε υπερβολική κατανάλωση ενέργειας και εξάντληση των φυσικών πόρων. Και πάλι λοιπόν αυτή είναι μια επιχειρηματολογία που πρέπει να μας οδηγήσει στη μείωση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, ιδίως μέσα στις ευρωπαϊκές τράπεζες επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που δίνει περίπου και η τράπεζα για ανασυγκρότηση και ανοικοδόμηση δίνει κάπως λιγότερο ποσό 9 δισεκατομμύρια εναντί 62 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ιδίως στις χώρες της Κεντροανατολικής Ευρώπης και οι δύο από αυτές τις τράπεζες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσουν τις οικονομίες και την ανάπτυξη της ενεργειακής τους υποδομής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τα τελευταία πέντε χρόνια δαπάνησε 62 δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα της ενέργειας. 34% από αυτά τα δισεκατομμύρια πήγανε για να υποστηρίξουν σχέδια που εμπλέκουν ορυκτά καύσιμα. 2 δισεκατομμύρια για τον άνθρακα. Αυτό είναι το συνολικό ποσό δανειοδότησης. Αν δούμε σε περιφερειακό επίπεδο τι γίνεται, βλέπουμε ότι στις νέες χώρες μέλη, Κεντροανατολική Ευρώπη, το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων, των σχεδίων ορεινών καυσίμων που υποστήριχε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν πολύ πιο υψηλό από ό,τι στις λεγόμενες χώρες της παλιάς Ευρώπης. Βλέπουμε και έξω από την Ευρώπη ότι τα σχέδια που έχουν ορυκτά καύσιμα παίρνουν περισσότερη δημόσια επιδότηση από ό,τι άλλα σχέδια. Και οι δύο τράπεζες κάθε πέντε χρόνια αναθεωρούν την ενεργειακή του πολιτική η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το κάνει εφέτος και μέχρι το καλοκαίρι εφέτος θα έχουν μια πρόταση για μια νέα ενεργειακή πολιτική που θα καθορίσει την στρατηγική δανειοδότησή του για τα επόμενα πέντε χρόνια. Και βλέποντα τι μακροχρόνιε προοπτικές είναι σαφές ότι δεν πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω ο άνθρακας μέσα στις ε, χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων. Περισσότερη υποστήριξη πρέπει να δοθεί στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στις ανανεώσιμες ενέργειες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης έχει μια έχουμε εδώ μια παρόμοια κατάσταση σε σχέση με τις δανειοδοτήσεις 48% μεταξύ 2006-2011 πήγανε στα ορυκτά καύσιμα, πολύ λιγότερο ήταν οι ανανεώσιμες ενέργειες και η ενεργειακή απόδοση. Και αυτή η τράπεζα το 2013 το καλοκαίρι θα αναθεωρήσει την πολιτική της και εκεί πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι για να υποστηρίζουν την, τα σχέδια παραγωγής ενέργειας από άνθρακα πρέπει να επιταχύνουμε τη μετάβαση στις ανανεώσιμες ενέργειες και γι' αυτό πρέπει να μπουν περισσότερα δημόσια κονδύλια στην αποδοτικότητα της ενέργειας και στις ανανεώσιμες ενέργειες. Μπορώ να σταματήσω εδώ λοιπόν. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ τα μάλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο. Κυρία Κάουτης, της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών, ευρωπαϊκών φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση την οποία μου απευθύνατε. Ε, ανήκω στην Ένωση Φωτοβολταϊκών Βιομηχανιών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά και θα σας μιλήσω για τις δυνατότητες στον τομέα της ανανεώσιμης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρώτον θα πω γιατί θα πρέπει η Ευρώπη να στοχεύσει σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο παραγωγής από ανανεώσιμες. Δεύτερον, ποιος ο ρόλος που μπορεί να παίξει το φυσικό αέριο και ο άνθρακα στη μεταβατική περίοδο και τέλος θα καταλήξω με ορισμένες ε, συστάσεις κατευθύνσεις από πλευράς μας. Γιατί η Ευρώπη θα πρέπει λοιπόν να στραφεί σε ένα σύστημα ανανεώσιμων πηγών. Νομίζω ότι και το οικονομικό επιχείρημα είναι σαφές. Είδαμε ότι οι τιμές των καυσίμων συστηματικά αυξάνονται στις τελευταίες δεκαετίες. Ακούσαμε επίσης, το είπε ο κ. Σκέλη, ότι οι εισαγωγές το 2011 καυσίμων ανήλθαν σε 388 δις. Δηλαδή ένα δις ημερησίως για το σύνολο της Ευρώπης. Ακόμα και όταν έχει αρχίσει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάζει τα λεγόμενα μη συμβατικά καύσιμα, οι προβλέψεις των ε, διεθνών οργανισμών προβλέπουν ότι ο λογαριασμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Ό,τι και να κάνουμε δηλαδή, αν παραμείνουμε στα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρισμού, θα αυξηθεί το κόστος. Αν εξετάσουμε τις ανανεώσιμες πηγές συγκριτικά βλέπουμε ότι η ανταγωνιστικότητά τους βελτιώνεται, μειώνονται το κόστη, έχουμε σημαντικές μειώσεις του κόστους με συστηματικούς ρυθμούς. Βλέπουμε ότι έχουμε συστήματα που φτάνουν σε μειώσεις μέχρι 32%. 15% τα τελευταία χρόνια, ένα πολύ σημαντικό βήμα και η αιωλική ενέργεια και η ηλιακή ενέργεια ξέρετε ότι δεν χρειάζεται ε, ορυκτές πηγές καυσίμων και θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε και τα εμπορικά ελλείμματα τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Βλέπετε εδώ τις, τους ιστούς της αράχνης βλέπετε τις διαφορετικές μορφές αντιμετώπισης της ανταγωνιστικότητας. Από τη μία βλέπετε την εξίσωση της δυναμικής σύγκρισης των δικτύων για οικιακή χρήση. Βλέπουμε εδώ ότι αν υπήρχαν συστήματα οικιακά από εναλλακτικές πηγές θα κατανάλωναν μόνο τα νοικοκυριά το 30% της ενέργειας που καταναλώνουν σήμερα. γιατί δεν θα έχουν ανάγκη να αγοράζουν τον ηλεκτρισμό τον οποίο αγοράζουν σήμερα. Αυτή η δυναμική εξίσωση λοιπόν το, σε σχέση με τη συμμετοχή στα δίκτυα βλέπουμε ότι διαφέρει από χώρα σε χώρα και μπορούν όμως σε διάφορες χώρες ε, να την πετύχουν αρκετά γρήγορα μέχρι το 14-15 στην Ιταλία και από το 15 με 18 στη Γαλλία. Ο δεύτερος ιστός ε, είναι μια σύγκριση του κόστους ε, της δικτύωσης και των εγκαταστάσεων με την χρήση 4.000 ωρών κατέτος γεννητριών από, που τα οποία, οι οποίες λειτουργούν με φυσικό αέριο και βλέπουμε ότι σε χώρες όπως η Ιταλία από το 12 μέχρι το 14 θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση ενώ σε άλλες χώρες από το 15 και μετά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα επιβληθούν από μόνες τους οι ανανεώσιμες πηγές και δεν θα συμβεί τίποτα περισσότερο. Όλα θα εξαρτηθούν από τις ρυθμίσεις τις νομικές και πολιτικές και υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που θα παίξουν ρόλο, αλλά αυτά σας δείχνουν ότι οι τιμές των ανανεώσιμων δεν είναι στα υψηλότατα επίπεδα, στα υπερβολικά επίπεδα τα οποία έχουν πάρα πολύ στο νου τους και είναι πάρα πολύ κοντά στις τιμές του ηλεκτρισμού έτσι όπως παράγεται σήμερα στην αγορά. Το θέμα δεν είναι μόνο ο οικονομικός παράγων, το θέμα είναι και τι περιβαλλοντικά ωφέλη έχουμε από τις ανανεώσιμες πηγές και εδώ είναι ιδιαίτερα πιστικά τα επιχειρήματα. Ακούσαμε για το χαμηλό ίχνος, όπως φαίνεται εδώ στο γράφημα. Βλέπετε όταν συγκρίνουμε τη, ζωή, τη διάρκεια ζωής μιας μονάδας ανάλογα με την πηγή με την οποία ε, παράγεται ο ηλεκτρισμός. Αριστερά βλέπετε το πετρέλαιο, τον άνθρακα, το φυσικό αέριο και δεξιά βλέπετε τις εναλλακτικές πηγές. Το θέμα δεν είναι μόνο βέβαια ο άνθρακας. Ξέρουμε ότι έχουν μειώσει εντελώς α, ε, οι ανανεώσιμες πηγές στην εκπομπή και άλλων α, ε, απειλητικών τοξικών όπως το μονοξίδιο του άνθρακα τα αζωτούχα, τα φιούχα, το μεθάνιο και το όζον. Επίσης μειωμένη κατανάλωση ε, υδάτινων πηγών, χαμηλότερη θερμική ε, μόλυνση κτλ. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι για να μπορέσει η Ευρώπη να έχει μια βιώσιμη και αηφόρο όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και οικονομική ενεργειακή πολιτική χρειάζεται να κινηθεί και προς τις ανανεώσιμες πηγές. Στον οδικό χάρτη για το 2050 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι τουλάχιστον το 50 με 70% των ανανεώσιμων θα απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι το 50. Στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού το 50% αυτό θα είναι πολύ ανώτερο το συστημικό κόστος των ανανεώσιμων δεν θα είναι υψηλότερο από το τι ισχύει σήμερα και από όλα τα άλλα σενάρια που ισχύουν σήμερα. Και όχι μόνο για τη δεκαετία του 50, του 2050, αλλά και για τις δεκαετίες οι οποίες μεσολαβούν. Εν πάση περιπτώσει όπως και να έχουν τα πράγματα τα κόστη θα αυξηθούν. Αλλά στην περίπτωση των ανανεώσιμων δεν θα αυξηθούν περισσότερο από ό,τι τα υπόλοιπα σενάρια. Τώρα, αν περάσουμε σε ένα ανανεώσιμο σύστημα, ποιος θα είναι ο ρόλος του άνθρακα και του φυσικού αερίου. Κοιτάξτε, πώς θα έχει ένα τέτοιο σύστημα, πώς θα είναι ένα τέτοιο σύστημα. Θα υπάρχει μια παραγωγή πιο αποκεντρωμένη, θα χαρακτηρίζεται από πολλαπλές ανανεώσιμες πηγές, άνεμος, ήλιος, αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μια μεγαλύτερη ευελιξία στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στην κατανάλωση φυσικά του ηλεκτρισμού, στις οποίες ανταποκρίνεται ο, ο τομέας. Τώρα, ακριβώς λόγω των διαφορών στην παραγωγή, απαιτείται μια περαιτέρω ευελιξία. Ο τομέας μπορεί με ένα σωστά διασυνδεδεμένο σύστημα να παράσχει την απαιτούμενη ευελιξία και μέσω της αποθήκευσης και μέσω της ελεγχόμενης διακύμανσης στην παραγωγή. Μία από τις πηγές ευελιξίας είναι τα ορυκτά συστήματα όπως το πετρέλαιο κτλ. και μπορεί να χρησιμοποιηθούν στις ενδιάμεσες φάσεις. Ποιος είναι ο ρόλος λοιπόν για τον άνθρακα και το φυσικό αέριο στην μεταβατική περίοδο. Εμείς δεν θα έχουμε αύριο την απόλυτη 100% χρήση των ανανεώσιμων πηγών. Τα ορυκτά καύσιμα θα παραμείνουν στο σύστημα, αλλά αυτά τα οποία θα παραμείνουν θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά και ευέλικτα. Σε σχέση με την ασφάλεια των συστημάτων, αυτό το οποίο βρίσκουμε σε μια μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, είδαμε ότι η ασφάλεια της προμήθειας ενέργειας στην Ευρώπη δεν θα είναι σημαντικό θέμα μέχρι το 2020. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει έτσι και αλλιώς στο σύστημα λόγω των διακυμάνσεων στη ζήτηση. Το 2020 θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα τα οποία να καλύψουν τις διαφορετικές διακυμάνσεις. Αυτά έχουν σχέση με τις διασυνδέσεις των συστημάτων, με την αποθήκευση της ενέργειας και την αποκεντρωμένη παραγωγή της ενέργειας. η σκέψη του να υπάρχουν μονάδες παραγωγής οι οποίες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο συνεχώς σε αιτήσια βάση χωρίς να ανταποκρίνονται και να αλλάζουν ανάλογα με τις διακυμάνχεις της ζήτησης είναι κάτι που δεν θα υπάρχει στο μέλλον. Τώρα, πώς μπορούν τα συστήματα από ορυκτά καύσιμα να λειτουργήσουν στις συνδυασμένες μορφές παραγωγής. Υπάρχουν διαφορές τεχνολογικές και οικονομικές ανάμεσα στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Ε, γενικότερα θα έλεγε κανείς ότι οι μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου είναι πιο ευέλικτες από τις μονάδες παραγωγής με άνθρακα. Ε, επίσης ε, Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες έτσι κι αλλιώς ευελιξίας, τις οποίες μπορείτε να δείτε στον προηγούμενο πίνακα. Λοιπόν, τώρα για τον ρόλο των καυσίμων αυτών στη μεταβατική περίοδο. Θα παίξουν ένα ρόλο λοιπόν, υπάρχουν πολλές επιλογές για να δώσουν οι παραδοσιακές αυτές μορφές παραγωγής την ευελιξία την οποία έχει ανάγκη το σύστημα. Κλείνοντα θα ήθελα να συνδέσω το θέμα με τους λεγόμενους capacity mechanisms, δηλαδή τις δυνατότητες δημιουργίας περαιτέρω δυναμικού και δυνατοτήτων. Σήμερα το πρωί υπόθηκε άλλωστε ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα απαιτηθούν έτσι ώστε να υπάρξουν νέες επενδύσεις και να υπάρξει και μεγαλύτερη ευελιξία. Εδώ υπάρχουν κάποια επιπλέον θέματα τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Σε πάρα πολλά τμήματα της Ευρώπης υπάρχει υπερπαραγωγή θα έλεγα και όχι έλλειψη παραγωγής. Είδαμε επίσης ότι οι νέες δυνατότητες παραγωγής στην Ευρώπη θα πρέπει να βασίζονται κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές, ενώ η συζήτηση που γίνεται επίσημα αφορά μόνο τα ορυκτά καύσιμα. Υπάρχει ο κίνδυνος επίσης υπονόμευσης της αγοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ακριβώς των δεσμευμένων επενδύσεων και των περιορισμών στην χρήση του άνθρακα. Έχουμε επίσης περαιτέρω δυναμικό ευελιξία στο σύστημα που παραμένει μη εκμεταλλεύσιμο. Θέματα διασύνδεσης, DSM, θέματα αποθήκευσης και τέλος Μπορούμε να δικαιολογήσουμε την υποστήριξη ε, των ε, επιδοτήσεων για να οριμάσουν οι τεχνολογίες οι οποίες αυτή τη στιγμή στηρίζονται. Τώρα τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς θα πρέπει να αναγεννήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα μέσα κλιματολογικής της πολιτικής. Είτε επισκευάζοντας το σύστημα ETS, είτε ε, εφαρμόζοντας νέα μέτρα όπως σαν παράδειγμα στον τομέα της παραγωγής νέες μελέτες. Θα πρέπει επίσης να τεθούν νέοι στόχοι για το 2030 για τις ανανεώσιμες πηγές, για το κλίμα και την αποδοτικότητα. Κοιτάξτε δεν έχω άλλο χρόνο, θα πρέπει να σταματήσω πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Λέει Πρόεδρος. Έχει το λόγο ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ένα θέμα το οποίο έχει ήδη συζητηθεί, το θέμα της αποθήκευσης της ενέργειας. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι το εφικτό αλλά υπάρχει κάτι το πιο σημαντικό που πρέπει να προηγηθεί. Πρέπει να διασφαλιστεί η διασύνδεση με υψηλή αποδυτικότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το υπερδίκτυο, το super grid. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε όλες τις μορφές παραγωγής σαν να ήταν μία όλες οι πηγές μαζί. Και έτσι θα πρέπει να υπάρξει και μία αντιστάθμιση στατιστική και των μορφών παραγωγής αιωλικής Αυτή η μεταφορά ηλεκτρισμού με υψηλή τάση μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την υδρολογική, υδροηλεκτρική παραγωγή για να αντισταθμίσουμε μια πιθανή έλλειψη παραγωγής από πλευράς αιωλικών πηγών ενέργειας. Μία άλλη δυνατότητα την οποία έχουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το φυσικό αέριο που έχει τις δικές, της δυνατότητες, τις δικές του δυνατότητες αποθήκευσης και που διασφαλίζει επίσης και μία πολύ μεγαλύτερη ευελιξία. Σας υπενθυμίζω την γερμανική εμπειρία μικρογεννητριών θα έλεγα με αποθήκευση θέρμανσης που μπορεί να παράγει ενέργεια ανάλογα με τις απαιτήσεις και τη ζήτηση του δικτύου και η θερμότητα αυτή η οποία έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε μας παρέχει θα έλεγα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να σκεφτούμε άλλες δυνατότητες όπως το υδρογόνο που πολλές φορές περιλαμβάνει περάσματα από τεχνολογίες χαμηλής αποδοτικότητας. Επίσης υπάρχουν ε, και κάποιες ε, δυνατότητες δημιουργίας εγκαταστάσεων άντλησης που και αυτές ε, μπορούν να μας δώσουν αποτελεσματικές δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το σύστημα με συνολικό τρόπο από τις τεχνολογίες οι οποίες έχουμε στη διάθεσή μας, είναι του χεριού μας θα έλεγα, μπορούμε χρησιμοποιώντας τες να προχωρήσουμε σε ένα εξορθολογισμό πολύ σημαντικό του ενεργειακού μας συστήματος. Και φωτοβολταϊκό που έχει μια καμπύλη θα έλεγα παραγωγής. Αυτή η καμπύλη παραγωγής είναι πάρα πολύ αντίστοιχη με τη ζήτηση των βιομηχανικών μονάδων. Είναι λοιπόν μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Έχουμε όλες τις γνώσεις που απαιτούνται και απλά θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να επενδύσουμε για να εξορθολογήσουμε το ενεργειακό μας σύστημα βελτιώνοντας την αποδοτικότητά του και μειώνοντας το περιβαλλοντικό του ίχνος. Ευχαριστώ συνάδελφε Πρόντι. Θα δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο Γκριμς. Να χαιρετήσω μια αντιπροσωπεία η οποία ήρθε. Βλέπω ότι είστε Ιταλοί, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το 4 στα ακουστικά σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πάντα κάνω μια πρόταση. Δεν πρέπει να καταδικάζουμε τον άνθρακα. Γιατί ο άνθρακας είναι απαραίτητος για τη ζωή. Δεν πρέπει να είναι αποδιοπεμπαίος ε, τράγος. Χρειαζόμαστε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών, όχι χαμηλής ε, κατανάλωσης άνθρακα. Βέβαια, το θέμα διαφέρει όταν περνάμε ε, στα ορυκτά. είναι μάλλον επιστημονική παρατήρηση. Η οικονομία χαμηλών εκπομπών. Ναι, έχετε δίκιο. Οι εκπομπές από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ χαμηλότερες από τις εκπομπές ε, από ρηκτά καύσιμα και οι εκπομπές ε, που προέρχονται από τον άνθρακα είναι υψηλότερες από αυτές που προκύπτουν από το φυσικό αέριο. Όμως να θυμάστε ότι με σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομέ μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές από τον άνθρακα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα κοινό παρανομαστή. Στην παρουσίασή σας επιβεβαιώσατε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτές εκλείουν ε, διοξιδίου του άνθρακα και εκπομπέ. Για τα φωτοβολταϊκά χρειάζεται η αύξηση ε, των εκπομπών. Όμως ε, η ενεργειακή ισορροπία είναι διαφορετική. Πριν από λίγο καιρό μιλούσαμε για τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαθεσιμότητα ή έλλειψη αυτής. Η, αποτελεί τροχοπέδι για την παραγωγή ενέργειας. Μιλώ εδώ για τα φωτοβολταϊκά που απαιτούν την χρήση σπάνιων γεών. Θέλω λοιπόν να βρούμε κοινού παρονομαστέ για τα φωτοβολτικά. Προφανώ απαιτείται ηλιακή ενέργεια, ήλιο. Πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ε, την ε, συνέχεια και την ασφάλεια της παραγωγής με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου μέσω της μικροπαραγωγής, Micro generation. Ε, σήμερα ολοκληρώνουμε τις διαπραγματεύσεις για τη μικροπαραγωγή. Έχω δει κάποιες ε, εγκαταστάσεις στην Πολωνία, πιλωτικές εγκαταστάσεις που δείχνουν πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα φωτοβολταϊκά, την ηλιακή ενέργεια με την τοπική μικροπαραγωγή βάση του φυσικού αερίου. Με 90% αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα κυρίε και κύριοι και αυτό είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα χάρη ε, στις τεχνικές παραμέτρους. Είναι λοιπόν ε, μια ε, συνέργεια που απαιτείται. Υπάρχουν και κάποια εμπόδια βέβαια ε, που αποτελούν τροχοπέδι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εγωιστικές ε, τάσεις σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο βιομηχανίας. Αναφέρατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αγοράζει πολλή ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, διαμορφώσει ικανότητα μετάδοσης ενέργειας ε, διπλάσιας δυναμικής ε, σε σχέση με τον όγκο της ενέργειας που πωλείται από τη Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 300 δις είναι προς το παρόν, αλλά έχουμε διαμορφώσει νέα ικανότητα μετάδοσης της ενέργειας, γιατί θέλουμε να, είμαστε, να αποκτήσουμε την ανεξαρτησία μας. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Ανανεώσιμε πηγές ενέργειας θα πρέπει να διαμορφωθούν ε, πρώτα απ' όλα στις περιοχές ε, που είναι φτωχέ σε ενέργεια. Όμως, στην πραγματικότητα, οι μεγάλε πολυεθνικέ ε, θέλουν να καπηλευθούν αυτές τις αγορές προς όφελό τους. Και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε κριτικά. Εφόσον ενώσιμες πηγές ενέργεια, υποτίθεται ότι θα δώσουν όθηση στις φτωχέ σε ενέργεια περιοχές, κυρίως τι αγροτικέ. αυτή η ενδυνάμοι ε, παραγωγή ενέργειας προσπαθούν ε, να δραστηριοποιηθούν, αλλά αποτυγχάνουν. Βεβαίω και θέλουμε να στηρίξουμε ε, τι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, αλλά χρειαζόμαστε και χρηματοδότηση. Και κάποιες φορές εκ των υστέρων αλλάζουν τα κριτήρια και καταργούνται τα κίνητρα, όπως έχω πει και προηγουμένως θα πρέπει να στραφούμε προς την εξέβραση συμβιβαστικής λύσης. Να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις προς την παραγωγή ενέργειας και τους ενεργειακούς πόρους. Ο εκπρόσωπος ε, της πολωνικής επιχείρησης ε, φυσικού αερίου και πετρελαίου είπε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την έρευνα στην ενεργειακή αποθήκευση που θεωρώ ότι θα διευκόλυνε την αποτελεσματική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων πηγών ενέργειας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήλπιζα ότι θα ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τις βασικές προκλήσεις. Βλέπουμε ότι το κόστος της βιομηχανίας αυξάνει, το κόστος της ενέργειας αυξάνεται, το κόστος ε, της στρατηγικής του 2050 διπλασιάζεται και δεν βλέπω να έχουμε καμία δυνατότητα να ελέγξουμε σε επίπεδο πολιτικής αυτές τις τάσεις, όπως φάνηκε και από τη συζήτηση για το ETS την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε κονδύλια για την κατεύθυνση αυτή. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. πρέπει να περάσουμε από την τιμολόγηση βασί πόρων σε μια πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένη βιομηχανία. Αλλιώς θα παραμείνει η βιομηχανία δεσμευμένη από τους ε, φυσικούς πόρους. Πώς θα το κάνουμε αυτό, αν δεν μπορούσαμε να το κάνουμε σε εποχές παχαίων αγελάδων, πώς θα το κάνουμε τώρα. Πώς θα εξασφαλίσουμε η κοινή γνώμη να μας υποστηρίξει προς την κατεύθυνση αυτή. Μ' άρεσαν και δύο παρουσιάσεις. Αλλά με οδήγησαν σε περισσότερες ανησυχίες. Ναι, τα χρειαζόμαστε όλα αυτά και ποιος θα τα πληρώσει. Θα μας υποστηρίξουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αν δεν θέλουν, τι θα κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πραγματικά ασθενής και ανεπαρκής η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ε, Τα χρήματα που παίρνουμε από τη βιομηχανία είναι κυρίως θέματα έρευνας και η έρευνα είναι από τους μεγαλύτερους χαμένους στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Η οπισθοφόρτηση αναφέρθηκε προηγουμένως. Αλλά είναι μόνο η δική μου χώρα που είπαν όχι να ξαναγυρίσουμε στα κρατικά μονοπόλια και να μην ε, προχωρήσουμε σε κοινοτομία Ή το κάνουν όλες οι χώρες. Τι θα κάνουμε λοιπόν αν δεν υπάρξει πρόοδος. Ε, ευχαριστώ. Ματσκίεβιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Η συζήτηση έχει αρχίσει να γίνεται πολωνοπολωνική. Όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι από τη χώρα μου έχουν πάρει το λόγο. Εγώ διάβασα πρόσφατα ότι αναζητούνται μέλη για την αποστολή στον Άρη. Είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει, θα έλεγα, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα και την έκπληξή μας κάθε φορά που αλλάζουν τα πράγματα. Όλοι όσοι πήραν το λόγο εδώ και κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας παράλληλα συμφωνούν ότι κάποιοι παγκόσμιοι παίκτες όπως η Νότια Αφρική, η Ινδία, η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείες επηρεάζουν κατά πολύ τα πράγματα και δυσκολεύουν την επίτευξη συμφωνίας στο πακέτο για το κλίμα. Το πρωτόκολλο στο Κιώτο ε, είχε μεν συμφωνηθεί πριν αρκετά χρόνια, αλλά δεν υπάρχει ενθουσιασμός ε, για περαιτέρω βήματα. Υπάρχουν ε, συνεχείς επίσης συζητήσεις για μετακινήσεις επιχειρήσεων, για διαφορετικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές και χώρες και συνεχείς συζητήσεις για χαμηλότερες πηγές ενέργειας σε διαφορετικά μέρη σαν βουλευτές θα πρέπει να μην ξεχνάμε ποιους αντιπροσωπεύουμε πάντως εμείς εδώ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια κοινή αγορά ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση της βιομηχανίας και την κατάσταση στον τομέα της απασχόλησης. Γιατί εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα. Θα πρέπει να αναζητήσουμε λοιπόν μια κάποια συμβιβαστική λύση να χρησιμοποιήσουμε όλες τις διαθέσιμες πηγές παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμες ή Υπάρχει κάποιος χρόνος και υπάρχει δυνατότητα σταδιακής προσπάθειας συνδυασμού ε, για να καταλήξουμε σε μια διαφορετική οικονομία της ενέργειας. Δεν μπορούμε βέβαια να αλλάξουμε βία την κατάσταση γιατί υπάρχουν απότομες διακυμάνσεις στην παραγωγή ενέργειας από Εναλλακτικέ πηγές. Πολλοί μίλησαν για την ευελιξία. Η ευελιξία είναι μια μαγική λέξη, η οποία πολλές φορές όμως αντικαθιστά τα πραγματικά επιχειρήματα. Οι Κινέζοι έχουν κάνει πάρα πολλά στον τομέα αυτό και αυτό το οποίο απαιτείται πάντως σε μας είναι να υπάρξει μια σταδιακή πρόοδος προς τη συνδυασμένη χρήση των τεχνολογιών όσο οριμάζουν οι τεχνολογίες και όσο ενσωματώνονται οι ανανεώσιμες πηγές στα παραδοσιακά δίκτυα, κάτι το οποίο σήμερα είναι προβληματικό. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τις ορυκτές πηγές που είναι διαθέσιμες, δεν θα καταστρέψουμε το σύστημα που υπάρχει. Ευχαριστώ η συνάδελφος Ήμπνερ. Ευχαριστώ κύριε, Πρόεδρε. ο κύριος, ο προηγούμενος ομιλητής, ο κύριος Τρίλινγκ μας έδωσε ορισμένα στοιχεία που με <clears throat> εξέπληξαν τα μάλα. Από πού τα βρήκατε αυτά τα στοιχεία, τις πληροφορίες για τα ορυκτά καύσιμα. Γιατί ένας άλλος ομιλητής έδωσε τελείως διαφορετικά στοιχεία. Είπε ότι τα ορυκτά καύσιμα, οι τιμές των ορεικτών καυσίμων καταραίουν, μειώνουν, μειώνονται. Και αυτό οδήγησε στους Γερμανούς να κατασκευάσουν σταθμούς καύσης άνθρακα. Και επίσης κάτι τέτοιο ισχύει και για τα ορυκτά καύσιμα και την, τις τιμές του στην Κίνα. Θα ήθελα να ξέρω από πού έρχονται οι δικές σας πηγές για τα στοιχεία. Πού, από πού τα αντλείτε αυτά τα στοιχεία. Ένα ακόμα ερώτημα. Είπατε ότι μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν πέσει μέχρι και 50% οι τιμές της ανανεώσιμης ενέργειας. Από πού παίρνετε αυτά τα στοιχεία. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει στη ζωή μου. Πολύ ενδιαφέρον είναι, αλλά μπορείτε να το τεκμηριώσετε από κάποιες αξιόπιστες πηγές. Δεν συμφωνώ να εφαρμόσουμε περιορισμούς στη βιομηχανία μας, επειδή δεν μπορέσαμε να εγκρίνουμε την μεταρρύθμιση του ETS που υποτίθεται δεν δουλεύει. Μια χαρά δουλεύει το ETS. <clears throat> Είναι ένας μηχανισμός που βασίζεται στην αγορά. Και το εισαγάγαμε εμείς οι ίδιοι. Λειτουργεί στην πράξη, μπορεί να μην μας ικανοποιούν τα αποτελέσματά του, αλλά αυτό είναι διαφορετικό θέμα. Θεωρήσαμε ότι το, τα έσοδα του ETS θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περισσότερη καινοτομία και τεχνολογίες εχμή. Κατάσταση στην αγορά όμω είναι όπως είναι και έχουν πέσει τιμέ άνθρακα. Αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το σύστημα που εισαγάγαμε πριν από 7 χρόνια. Τονίσαμε ότι πρέπει να υπάρχει μια αξιοπιστία και μια προβλεψιμότητα που θα ευνοήσει τα κίνητρα και τις επενδύσεις. Θα ε, μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε ένα σύστημα που βασίζεται στην αγορά και το οποίο δουλεύει θαυμάσια. Δεν πρέπει λοιπόν να διαδίδεται ε, παραπλανητικές πληροφορίες. Μην λέτε το σύστημα δεν δουλεύει, το συζητήσαμε στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Είπαμε ότι μπορεί να, μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικό όσο θέλαμε, αλλά δουλεύει. Και όταν μας δίνετε δεδομένα θα πρέπει να βασίζονται σε ανεξάρτητες πηγές. Δεν μπορούμε να ακούμε στοιχεία που είναι αντιφατικά. Κλείσαμε λοιπόν τον κύκλο των παρεμβάσεων. Θα πρέπει να απαντήσουν οι εισηγητές μας. Τρίλινγκ. Thank you very much. I Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σχόλια και ιδέες που ακούστηκαν. Βλέποντας ε, την ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς, ε, τις επενδύσεις ε, στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, στα ΕΦΗ, e, δίκτυα για μακρινές αποστάσεις, αλλά και για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία και η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη ίσως να ήταν μια, ένας τρόπος ε, συμπλήρωσης αυτού του κενού επενδύσεων. Καλή ιδέα ήταν επίσης ε, το να βασιστούμε, να επικεντρωθούμε ε, σε μικρής κλίμακας ε, προσπάθειες και να δούμε τι είδους ενεργειακοί πόροι υπάρχουν εκεί, αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας και ενσωμάτωση διαφόρων τρόπων και μεθόδων και μέτρων. Αναφέρθηκε η έλλειψη ορισμένων ενεργειακών πόρων και επιστρέφω στο ζήτημα της, του θεματολογίου για το 2050, το ζήτημα της ενεργειακής ανταγωνιστικότητας. Τι πρέπει να προσπαθήσουμε, την απόλυτη αποσύνδεση της, των οικονομικών εξελίξεων και της αξιοποίηση ε, φυσικών πόρων. Επειδή είναι ε, σπάνιοι αυτοί οι πόροι, είναι πεπερασμένοι, δεν είναι θέμα ανταγωνιστικότητας λοιπόν πώς οι ευρωπαϊκές οικονομίες αλλά και παγκοσμίως μπορούν να επιβιώσουν όταν οικοδομούν τις οικονομικές τους δραστηριότητες και τις βασίζουν σε πεπερασμένους ενεργειακούς πόρους που συνεχώς μειώνονται. Πρώτον λοιπόν απαιτείται εδώ η, η αποθήκευση ενέργειας και εδώ συμφωνούμε όλοι. Και αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο για το ETS, το σύστημα εμπορίας εκπομπών, σκοπός ήταν η μείωση των ε, αερίων του θερμοκηπίου. Δεν δημιουργήθηκε για να δημιουργηθεί μια αγορά το ETS. Από αυτή την άποψη λοιπόν πρέπει ε, να επικρίνουμε την ιδέα ότι το δικαίωμα ε, ρήπανσης ε, του περιβάλλοντος πρέπει να τη χάνει εμπορίας μέσα στην αγορά και αν αποτύχει αυτή η αγορά ακόμα και αν αποτύχει, παραμένει η σωστή προσέγγιση. Πρέπει λοιπόν να δούμε τις ε, μακροπρόθεσμες εξελίξεις. Το 2050 υπάρχουν σαφείς στόχοι για τότε. Αποφάσεις για τις επενδύσεις στρατηγικές θα πρέπει να λεφθούν τώρα. Και επαναλαμβάνω δημόσια οικονομική και ρυθμιστική στήριξη που θα μας βοηθήσει να ε, φύγουμε από τα ρευστά καύσιμα και να ε, κινηθούμε προς μια οικονομία ε, χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα και εκπομπών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τίς. Ευχαριστώ να αντιδράσω σε κάποια από τα σημεία που τέθηκαν. Για τον κύριο Πρόντι και τη διασύνδεση. Θα συμφωνήσω μαζί του ότι το δίκτυο, το σύστημα των δικτύων είναι βασικό. Και για να αντισταθμιστούν οι διακυμάνσεις ανάμεσα στις περιοχές, και αυτό έχει σημασία ιδιαίτερα στην αιωλική, αλλά και στην φωτοβολταϊκή. Να ενισχυθούν τα συστήματα λοιπόν διανομής, και να υπάρξει δυνατότητα εφιούς διαχείρισης των συστημάτων. Και έρχομαι εδώ τώρα στο σημείο το οποίο τέθηκε για τις διακυμάνσεις οι οποίες αφορούν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες. Στα φωτοβολταϊκά οι αλλαγές δεν είναι πάρα πολύ βίαιες και είναι γενικότερα προβλέψιμες θα έλεγα σε μικρό χρονικό διάστημα. Το αν αυτές οι διακυμάνσεις μπορεί να αντιμετωπιστούν δεν τίθεται. Φυσικά και μπορούν. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις. Η πρόκληση είναι να βρούμε ποιες από τις λύσεις αυτές είναι οι πλέον θα έλεγα κατάλληλες και οι πλέον χαμηλού κόστους για να τις προωθήσουμε ανάλογα και να κάνουμε επιλογές. Είναι σαφές όμως ότι ε, ένα μίξ σωστής διαχείρισης του δικτύου, σωστών αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής και σωστής αποθήκευσης της ενέργειας θα είναι η λύση. Το θέμα είναι τι βάρος θα έχουν ο κάθε ένας από τους παραγόντες αυτούς. Σχετικά με τα φωτοβολταϊκά. Υπάρχουν κάποιες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται αν δείτε τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται δεν είναι πάρα πολύ υψηλέ σε σχέση με άλλους τομείς. Και τα καλά νέα είναι ότι τα συστήματα αυτά μπορεί να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Έχουμε δημιουργήσει κάποια προγράμματα έρευνας που προωθούν αυτή τη λύση. Ακούστηκε επίσης ότι η Ευρώπη δεν είναι απομονωμένη και ότι υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες θα πρέπει να λυθούν υπόψη. Σε μια εβδομάδα εμείς ε, θα εκδώσουμε τις προοπτικές μας τις μακροπρόθεσες για τη χρήση της ενέργειας. ενέργειας. Θα δούμε ότι η αγορά δεν συγκεντρώνεται αποκλειστικά στην Ευρώπη. Οι χώρες οι οποίες πρωτοπορούν είναι η Ιαπωνία, η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείες, και το θέμα δεν είναι να κάνει βήματα η Ευρώπη όταν οι άλλες δεν κάνουν. Το θέμα είναι η Ευρώπη να κρατήσει το πλεονέκτημα το συγκριτικό το οποίο έχει και να μην μείνει πολύ πίσω πλέον από τους άλλους. Και τέλος για την κυρία Χιμπνερ. Θέσατε δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά τις τιμές των καυσίμων των ορυκτών. Εγώ βασίστηκα στις προοπτικές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας έχει υπάρξει μείωση επίσης ε, του άνθρακα λόγω της πτώσης της ζήτησης του άνθρακα. Παρ' όλα αυτά η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προβλέπει ότι το κόστος ενέργειας για την Ευρώπη θα αυξηθεί. Και για τη μείωση στις ανανεώσιμες σας είπα ότι έχει μειωθεί κατά 15% το κόστος, 50% ε, το κόστος των φωτοβολταϊκών τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτά θα ε, μπορέσετε να τα ελέγξετε επίσης και μέσω των στατιστικών που έχουμε από τα ETS. Μπορείτε επίσης τα στοιχεία αυτά και στα τέλη τα οποία πληρώνονται για την παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Αν δείτε τα τιμολόγια τα οποία ε, πληρωνόντουσαν πριν 7%, 50%, ανά κιλοβατόρα ήταν 70 ε, σέντ του ευρώ ενώ τώρα είναι 15 με 30. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Λέβενστάιν από την προηγούμενη στρογγυλή τράπεζα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αντιμετωπίσω ένα σημαντικό θέμα, μια πρόταση η οποία διατυπώθηκε εδώ, ότι τα ορυκτά καύσιμα θα μας δώσουν μεγαλύτερη ευκαμψία μέχρι το 2020 και με τον τρόπο αυτό μπορούν να υποστηρίξουν την, την ε, χρήση ανανεώσιμων ενεργειών που είναι αστάθμητες σε σχέση με, τον, με το ύψος της παραγωγής ενέργειας. Αλλά πρέπει να ξεχάσουμε ότι όλα, όλη η, η εγκατάσταση σταθμού που έχει γίνει είναι για να επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα τέλη χρήσης του δικτύου ενεργείας για πρόσβαση στο δίκτυο. Πώς θα εξασφαλίσουμε λοιπόν τη βιωσιμότητα όλων αυτών των ε, νέων επενδύσεων όταν δεν έχουμε μια επαρκή αγορά. Υπάρχουν και πρόσθετες πηγές κόστους που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Εντάξει, λέει Νομίζω ότι μπορώ τώρα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Πάλι, κύριε Χίμπνερ, πάλι, 30 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ. Θα σας ευχαριστήσω και πάλι κύριε Πρόεδρε. Μόνο μία παρατήρηση. Αναφέρομαι σε αυτά που είπε η Επίτροπος κυρία Χέντεγκαρτ. 20% μείωση του διοξιδίου του άνθρακος δεν μπορεί να επιτευχθεί μέχρι το 2018. Ας μην είναι παραπλανητικά αυτά που λέτε. Υπάρχει ένας μηχανισμός που βασίζεται στην αγορά για το ETS. Άλλαξε στόχο και τη μείωση των εκπομπών και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει αυτά να μειώσουμε τις εκπομπές. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Ο κύριος Μοράλτ. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι δύσκολο να συνοψίσει κανείς ε, τα συμπεράσματα αυτής της δημοσίου ακρόασης σε μερικές ε, προτάσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που διοργάνωσε αυτή την ακρόαση. Νομίζω ότι ακούσαμε πολλά και ενδιαφέροντα για δύο από τους ε, τομείς. Και μετά βέβαια είχαμε και τα φωτοβολταϊκά εκ μέρους των ανάσωμα πηγών ενέργειας. Όλα αυτά μας έδειξαν πόσο περίπλοκαν όλα αυτά τα ζητήματα δείξαμε πολλά ανοιχτά θέματα. Υπήρξαν και κάποιες υπόνοιες ε, ε, για στοιχεία που απαιτείται μεγαλύτερη διερεύνηση και εμβάθυνση, για παράδειγμα για τις νέες τεχνολογίες, περισσότερη έρευνα, καινοτόμα προϊόντα. Και η συζήτηση περιστρέφει γύρω από το θέμα της ε, οργάνωσης της αποθήκευσης ενέργειας, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποιες ε, πηγές ενέργειας και να μετατρέψουμε τη μία μορφή σε άλλη. Σημαντικά ζητήματα όλα αυτά. Κάτι άλλο που ανέκυψε σε όλες τις ε, παρεμβάσεις ήταν η ανάγκη μαζικών επενδύσεων στις υποδομές τα σημεία σύνδεσης επίσης αναφέρθηκαν. Όλα αυτά τα μεμονωμένα ζητήματα, τα επιμέρους ζητήματα, κατά τη γνώμη μου πρέπει να τα εξετάσουμε στο ευρύτερο πλαίσιο ε, της ευρωπαϊκής ε, ενεργειακής και περιβαλλοντολογικής ε, πολιτικής. Και αυτό είναι, ήταν και το βασικό ε, και πρώτο σημείο της μέσης διάταξης σήμερα που αφορούσε την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Αυτό συγκρατώ και εγώ από τη σημερινή συζήτηση, η βάση περαιτέρω εξέλιξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ δεν ε, ε, βρίσκομαι σε αυτόν τον τομέα πολιτικής εδώ και πολύ καιρό. Την 1η Απριλίου ξεκίνησα. Βλέπω όμως μια σαφή τάση για ισχυρότερο κατακαιρματισμό ε, των αγορών παρά για μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Θεωρώ λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή αλλά και η Βιομηχανία πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιστρέψουμε αυτή την τάση και να κινηθούμε προς την ολοκλήρωση. Και εδώ οι ευθύνε είναι ξεκάθαρες. Η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πιέσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ε, το νομικό πλαίσιο που βρίσκεται σε ισχύ και μόνο όταν συμβεί αυτό μπορούμε να περάσουμε στην υλοποίηση όλων αυτών ε, που συζητήσαμε σήμερα, τότε θα βρουν τη θέση που τους αξίζει. Γιατί όσο δεν έχουμε υλοποιήσει αυτά που ε, έχουμε θεσπίσει, όλη αυτή η συζήτηση, δεν θα πω ότι δεν έχει νόημα, αλλά δεν θα βρει την κατάλληλη θέση ε, στην συνολική ενεργειακή και περιβαλλοντολογική πολιτική μας. Είναι λοιπόν προϋπόθεση για να επιτύχουμε αυτό που είχαμε δεσμευθεί για την ολοκλήρωση της ενεργικής αγοράς μέχρι το 2014, να το πράξουμε λοιπόν και μετά έχουμε τον επόμενο στόχο, το πλαίσιο για το 2030. Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ε, πράσινη βίβλο για δημόσια διαβούλευση και συνιστώ ε, σε όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ενεργά. Σε αυτό το διάλογο λοιπόν θα επανέλθουν όλα αυτά τα ζητήματα που ακούσαμε σήμερα. Στο τέλος, ακούσαμε τις αγορές ικανοτήτων, capacity markets. Δεν μπορούμε να έχουμε μια κρόαση μόνο για αυτό το θέμα, γιατί είναι ιδιαίτερα ακαθόδης ζήτημα. Ακούσαμε ότι το ETS ε, λειτουργεί μια χαρά όσο έχει και αυτό μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Συμφωνώ μαζί σας ότι ο πρωταρχικός μας ε, στόχος επετεύχθη από το ETS. Και μπορώ να σας πω ότι το 2020 θα έχουμε ξεπεράσει το στόχο μας κατά 0,9% κατά πάσα πιθανότητα. Τα υπόλοιπα αυτά ζητήματα λοιπόν έχουν τεθεί επιτάπητος δεν πρέπει να χάνουμε την προοπτική, να εξετάζουμε το συνολικό πλαίσιο, το οποίο για μένα είναι η κοινή ολοκληρωμένη αγορά ενέργεια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν τους εισηγητές μας, ευχαριστώ τους συναδέλφους που ήταν παρόντες. Εμείς θα συνεχίσουμε στις 3 το απόγευμα. Διακόπτουμε.